Okay. Μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση ελπίζοντας ότι θα αυξηθεί ο αριθμός των ατόμων που συμμετέχουν. Καταρχήν λοιπόν ερχόμαστε στην ημερήσια διάταξη. Θα ήθελα να σας πω ότι το σημείο 8 της ημερήσιας διάταξης ε, δηλαδή η συζήτηση με την Επίτροπο Κάθριν Άστον θα γίνει στις 10.30 και ε, ακριβώ μετά θα κάνουμε μια πάρα πολύ ε, σύντομη συνεδρίαση των συντονιστών και στο τέλος θα κάνουμε το αποχαιρετιστήριό μας, δηλαδή θα πιούμε ένα ποτήρι διότι τελικά είναι σήμερα η τελευταία συνεδρίασή μας ε, καθότι ολοκληρώνεται η περίοδος νομοθετικής θητείας. Εάν λοιπόν δεν έχετε παρατηρήσεις για την ημερήσια διάταξη και δεν βλέπω κάτι τέτοιο, ε, θεωρώ ότι έχει υιοθετηθεί. Και τώρα ερχόμαστε στο δεύτερο θέμα της ημερήσεως διαταξής, δηλαδή της ανακοινώσης του Προέδρου. Καταρχήν θα ήθελα να χαιρετήσω τον ε, πρεσβευτή της Κολομβίας ο οποίος ενδιαφέρεται ιδιαίτερως για το θέμα 7 το οποίο θα συζητήσουμε αργότερα. Ε, ανακοινώσεις του Προέδρου. Καταρχήν ε, πρέπει όταν μιλάτε επειδή ε, υπάρχει αναμετάδοση στην τηλεόραση να, να ε, πατάτε το κουμπί του μικροφόνου σας διαφορετικά δεν σας βλέπει η κάμερα. Επίσης εις τον ε, ε, κατάλογό σας υπάρχουν όλες οι επιστολές τις οποίες έχουμε αποστείλει ε, ο κατάλογος τουλάχιστον οπότε αν κάποιος θέλει να λάβει μία από αυτές τις επιστολές παρακαλείτε να απευθυνθεί στη γραμματεία για να του αποσταλεί επειδή σήμερα είναι η τελευταία μας συνεδρίαση θα ήθελα να υποφεληθώ της ευκαιρίας για να ευχαριστήσω όλους για τα δυόμιση χρόνια πολύ εντατικής, ε, ε, πολύ αποτελεσματικής και καρποφόρας ε, συνεδρία ε, ε, είχαμε δηλαδή πολύ ενδιαφέρουσες συνεδριάσεις της Επιτροπής ταξίδια θέλω να ευχαριστήσω και τους διερμηνείς οι οποίοι μας βοήθησαν και συνέβαλαν εις την κατανόηση παρόλο που περνούσαμε, ξεπερνούσαμε πάντοτε το ωράριό μας. Θέλω να ευχαριστήσω τη Γραμματεία. Είχαμε θαυμάσια συνεργασία, τουλάχιστον αυτήν την δικιά μου άποψη. Δεν ξέρω εσείς πώς το αξιολογείτε. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω όλους τους πολιτικούς συντονιστές, τους αρχηγούς των αντιπροσωπιών και όλους αυτούς οι οποίοι συμμετείχαν πάντοτε στις συνεδριάσεις μας και παρακολούθησαν τα θέματα που σας ενδιέφεραν στις, ε, στα διάφορα θεσμικά όργανα, στις ε, πρεσβείες και ε, σε όλους αυτούς οι οποίοι κατήρτισαν μελέτες πιστεύω ότι σαν Επιτροπή μπορούμε να θεωρηθούμε ότι είμαστε ικανοποιημένοι ε, διότι έγιναν όλα αυτά τα οποία επιθυμούσαμε και επιπλέον η πολιτική μπόρεσε ε, να ε, παρουσιαστεί καλύτερα στο Κοινοβούλιο. Θέλω όμως να σας διαβάσω μία επιστολή την οποία ε, γράψαμε χθες το βράδυ. Όταν ακούσετε την ανάγνωση θα καταλάβετε περί τίνος πρόκειται και ε, σήμερα ε, θα ήθελα να την αποστείλω τους συναδέλφους κατά τρόπον ώστε να συζητηθούν τα θέματα αυτά στις πολιτικές ομάδες διότι δηλαδή ενδέχεται την Τετάρτη να έχουμε μία ψηφοφορία επ' αυτού του θέματος στο Στρασβούργο και θα παρακαλούσα για την στήριξή σας. Η επιστολή είναι αγγλικά και θα, προσπαθήσω να το διαβάσω τουλάχιστον κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσει να καταγραφεί στα πρακτικά. Απευθύνεται στον κύριο Πέτερινγκ. Κύριε Πρόεδρε, το ψήφισμα το οποίο ε, υιοθετήθηκε στην Ολομέλεια στις 25 Μαρτίου για τις σχέσεις με τις χώρες ΑΚΕ έχει ε, την ε, παραπομπή στις συζητήσεις οι οποίες πρέπει να γίνονται από τις αρμόδιες επιτροπές και έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τις συμφωνίες οικονομικής συνεργασίας και ε, θα περιλαμβάνονται και στις ε, συμφωνίες οι οποίες θα ολοκληρωθούν. Η παράγραφος λέγει ότι θεωρεί ότι είναι σημαντικό η εφαρμογή των συμφωνισμών εταιρική σχέσεως να υπόκεινται σε ένα σύστημα παρακολούθησης η οποία θα οργανώνεται από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή με τη συμμετοχή των μελών της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και Επιτροπής Επιτροπής Αναπτύξεως για να εξασφαλιστεί η ισορροπία ε, σε όλα τα θέματα, δηλαδή στις ε, πολιτικές εμπορίου και ανάπτυξης. Θα πρέπει η Επιτροπή να αναβαθμιστεί και να συντονιστεί με την Κοινοβουλευτική Συνέλευση των χωρών και. Άκουσα ότι η και πληροφορήθηκα ότι στην σημερινή συνάντηση προβλέπεται ένας κατάλογος για τις διακοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες στις στα διάφορα θεσμικά όργανα. Αυτό ε, το κείμενο όμως ε, είναι αντίθετο στην ψηφοφορία που υιοθετήθηκε στην Ολομέλεια στις 25 Μαρτίου 2000 που αναφέρεται σαφώς και αναθέτει το ρόλο παρακολουθήσεως του Διεθνούς Εμπορίου εις ε, την αρμόδια επιτροπή και ε, εις ε, την επιτροπή συνεργασίας με τις χώρες ΑΚΕ. Θα πρέπει λοιπόν αυτό να ε, αναφέρεται σε αυτά τα θέματα και ε, ε, υπογράφω Helmut Μάρκοφ. Δεν βλέπω να υπάρχουν σχόλια. Οπότε μπορούμε να προχωρήσουμε στο τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης και θα επιθυμούσα να σας ανακοινώσω αλλά θα μιλήσω γερμανικά νομίζω καλύτερα ότι τα πρακτικά της, ε, της, των της συναντήσεως 16 Μαρτίου 2009 έχουν διανεμηθεί και ισχύει η ίδια διαδικασία. Δηλαδή αν μέχρι σήμερα το βράδυ δεν υπάρχουν αντιρρήσεις θεωρείται ότι έχουν υιοθετηθεί. Και έτσι περνάμε στο σημείο 4 το οποίο αναφέρεται στα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής της 24-25 Φεβρουαρίου, 5 Μαρτίου Μαρτίου και 16 Μαρτίου και ε, εάν δεν υπάρξουν αντιδράσεις μέχρι το τέλος της συνεδριάσεως θεωρούνται ότι έχουν υιοθετηθεί. Ερχόμαστε τώρα στο πέμπτο θέμα, εμπόριο πρώτων υλών. Όπως θυμάστε όλοι, το 2008 είχαμε καταρτήσει μία έκθεση κατά πρωτοβουλία της Επιτροπής μας που είχε αναλυφθεί από τον συνάδελφο Γιάννης Χόλμ και τώρα έχουμε την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις πρώτες ύλες. Όπως ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά πολύ εξαρτάται από την εισαγωγή πρώτων υλών και όταν κοιτάμε το έγγραφο αυτό μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι υπάρχουν τρία βασικά σημεία στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δηλαδή καταρχήν η επιθυμία να έχουμε τις ίδιες προσβάσεις προς τις πρώτες ύλες όπως και όλες, ε, όλοι οι άλλοι ανταγωνιστές μας. Δεύτερον, να μπορούμε κατά προτεραιότητα να έχουμε μία αηφόρο παράδοση και διαρκή παράδοση πρώτων υλών που να καλύπτουν τις ανάγκες μας και ότι η αποτελεσματικότητα ή στο θέμα της ανακύκλωσης των πρώτων υλών πρέπει να βελτιωθεί και ε, θα πρέπει συγχρόνως να μειώσουμε την κατανάλωση πρώτων ηρών. Εφόσον λοιπόν είναι εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία μπορεί να μας διευκρινίσει ακόμη την ανακοίνωση ε, θα δώσω το λόγο ή στην κυρία Μαντλέν Ντελίνκα και μετά στους συναδέλφους. Άρα η Επιτροπή έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ χρήσιμη αυτή η εισαγωγή. Χαίρομαι ιδιαίτερος που βρίσκομαι στην Επιτροπή σας. Όπως είπατε, μετά το ψήφισμα που υιοθέτησε πέρυσι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μετά την έκθεση αυτή, πολλές δραστηριότητε αναλύθησαν και πολλά ψηφίσματα που επιστέγασμά τους ήταν η ανακοίνωση που έχετε αναχείρας. Όπως είπατε, η ανακοίνωση αυτή ξεπερνά κατά πολύ τον τομέα του εμπορίου. Βέβαια το εμπόριο διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο παγκοσμίω. Αλλά το έγγραφο αυτό είναι ευρύτερο. Θα σας κάνω μία σύντομη παρουσίαση της ανακοίνωσης και μετά θα σας αναφέρω τις στρατηγικές εμπορίου, το σχέδιο δράσης, τις μελλοντικές προοπτικές και είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω στις απορίες σας. Εν αγωγής, Ήθελα να πω, όπως είπατε και εσείς, ότι ήταν ε, σαφής ο στόχος της ανακοίνωσης και τα κίνητρά της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξαρτάται ε, από την ε, εισαγωγή στρατηγικών πρώτων που υπάγονται σε στρέβλωση ανταγωνισμού πολλές φορές και το θέμα της εξόριξης αντιμετωπίζει συνθήκες ανταγωνισμού πολλές φορές όχι ιδιαίτερα θεμητού και υπάρχει ανάγκη για όλο και μια πιο ολοκληρωμένη αντίδραση και προσέγγιση, όπως πρότεινε το Συμβούλιο ήδη από το Μάιο του 2007. Για μία ανάλυση και τα προτινόμενα μέτρα ισχύουν και σε άλλα μη ενεργειακά υλικά, μη ενεργειακές πρώτες Η ανάλυση της ε, προσφοράς και της ζήτησης δείχνει ότι περάσαμε από μια εποχή αυτάρκειας σε μια εποχή μεγάλης εξάρτησης. Χρειαζόμαστε και πρωτογενή και δευτερογενή ε, πρώτε, ε, υλικά και δευτερογενείς και ε, πρώτες που είναι εξαιρετικά σημαντικές. Υπήρξαν σημαντικές αλλαγές και στις παγκόσμιες αγορές, στα χαρακτηριστικά τους και μία έρευνα που έγινε, μία απογραφή κατά τη διάρκεια του 2007 έδειξαν ότι υπήρχαν ε, σε 400 περίπου πρώτες ύλες 450 ε, περιορισμοί εξαγωγικοί και τα τελευταία δύο χρόνια έδειξαν οι μελέτες του ΩΣΑ ότι τέτοια μέτρα και τέτοιοι περιορισμοί έχουν πολλαπλασιαστεί. Επίσης ε, υπάρχουν στρατηγικές για προνομιακή πρόσβαση σε πρώτες ύλες σε ολόκληρο τον κόσμο. 50% των βασικών κοιτασμάτων ε, ορυκτού πλούτου βρίσκονται σε χώρες με χαμηλά εισοδήματα. Θέλουμε λοιπόν μια πιο ολοκληρωμένη στρατηγική και ήδη επισημάνεται τους τρεις πυλώνες κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα πρέπει να εξασφαλίσουμε πρόσβαση σε πρώτες ύλες ε, στις διεθνείς αγορές υπό ίσους όρους όπως και όπως για τους υπόλοιπους ανταγωνιστές μας. Επίσης θέλουμε ένα πλαίσιο με ισότιμους όρους ε, για βιώσιμη παροχή πρώτων υλών με εσωτερικό προσανατολισμό και επίση πρέπει να ενισχύσουμε τη συνολική αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα και να προωθήσουμε την ανακύκλωση για να μειώσουμε τη χρήση πρωτογενών ε, πρώτων υλών και να... την εξάρτησή μας από αυτές. Εγώ θα αναφερθώ στα βασικά στοιχεία του πρώτου πυλώνα επίκεντρό του είναι το εμπόριο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του επισήμανε πολλά από τα στοιχεία αυτά και εμά μα ενδιαφέρει το εμπόριο, το παγκόσμιο εμπόριο, αλλά το ανέφερε και σε άλλους τομεί. σε άλλα σημεία. μα ενδιαφέρει επίση το θέμα της ανάπτυξη και της βιωσιμότητα. και θα σα εξηγήσω πώ συμπεριλάβαμε και αυτά τα στοιχεία στην ανακοίνωσή μα. Η εμπορική μας στρατηγική είναι πολύ σχεδής. Καταρχήν, ε, τους τελευταίους μήνες ε, το θέμα αυτό πέρασε σε δεύτερη μοίρα, γιατί στο επίκεντρο των ανησυχιών μας βρέθηκε χρηματοπιστωτική κρίση. Και φυσικά το θέμα της πρόσβασης σε πρώτες ύλες είναι ένα μακροπρόθεσμο θέμα και δεν ε, μπορεί να τύχει άμεσης λύσης. Βέβαια, πρόθεσμα, οι τιμέ μπορεί να έχουν χαμηλώσει, αλλά στρεβλώσεις ανταγωνισμού υπάρχουν και επηρεάζουν ε, τις ευρωπαϊκές εταιρείε. Ποιοι είναι οι στόχοι τώρα για την εμπορική μας στρατηγική. Θέλουμε καταρχήν να αντιμετωπίσουμε τις, ε, τους περιορισμούς στην πρόσβαση που επιβάλλουν οι τρίτες χώρες. και θέλουμε κυρίως να χτυπήσουμε μέτρα που δεν ε, είναι νόμιμα και θεμητά που δεν δικαιολογούνται δηλαδή από αναπτυξιακά και περιβαλλοντικά κριτήρια. Επιπλέον αναλύουμε κάποια μέτρα που ε, θέτουν σε κίνδυνο τη συνεχή παροχή πρώτων υλών ε, από, την, από τις οποίες είναι εξαρτημένη η Ευρωπαϊκή Ένωση ή στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό μεταξύ των ευρωπαϊκών εταιριών και των παρόχων τους προμηθευτών τους από τρίτες χώρες. Η πρόκληση είναι τεράστια και απορρέει από το γεγονό ότι όπω σα είπα δεν υπάρχει μια θαυματουργή λύση άμεση αντίδραση. Χρειαζόμαστε συζητήσεις σε διμερή και πολυμερή επίπεδα, όπω φάνηκε και από τη δυσχέρεια των παγκόσμιων ε, εμπορικών διαπραγματεύσεων. Αλλά θέλουμε μια συνεκτική εμπορική πολιτική με πολλές πτυχές. Η στρατηγική του εμπορίου στηρίζεται σε τρεις πυλώνες που είναι διαφορετικοί μεταξύ τους. Ο πρώτος πυλώνας αφορά τις διαπραγματεύσεις και σε πολυμερές αλλά και σε διμερές επίπεδο προκειμένου να θεσπίσουμε κάποιους κανόνες. Στην Παγκόσμια Οργάνωση Εμπορίου μιλούμε για εξαγωγικούς δασμούς, για περιορισμούς εξαγωγικούς, στο σύστημα τιμολόγησης, τις επιδοτήσεις, τον ανταγωνισμό και τις επενδύσεις. Λαμβάνοντας φυσικά υπόψη και τις απαραίτητες εξαιρέσεις. Το ίδιο ισχύει και για τις διμερείς διαπραγματεύσεις. Εκεί βέβαια έχουμε περισσότερες ευκαιρίες ε, θέσπισης τέτοιων κανόνων, γιατί εκεί ε, το εύρος των εμπορικών διαπραγματεύσεων είναι μεγαλύτερο. Έχουμε διάφορες εμπορικές συμφωνίες με χώρες Κεντρικής Αμερικής, την Κορέα, την Ινδία και σε όλες αυτές τις διαπραγματεύσεις ε, το θέμα των κανόνων βρίσκεται στο επίκεντρο. Υπάρχει και δεύτερος πυλώνας που αφορά την ε, εφαρμογή και την ανάλυση αυτών των περιορισμών. Μερικές φορές υπάρχει κατάφορη καταστρατήγηση των διεθνών κανόνων. Υπάρχει ε, ένας μηχανισμός διακανονισμού των διαφορών και στην Παγκόσμια Οργάνωση Εμπορίου, αλλά προβλέπεται και από διμέρισμα συμφωνίες. Δίνουμε προτεραιότητα και στις εταιρικέ σχέσεις για την πρόσβαση στην αγορά. Θέλουμε να βελτιώσουμε τις προτεραιότητες μας εκεί και να συνεργαστούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να συνεργαστεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τις εθνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Τρίτος πυλώνας είναι ο διάλογος. Και διμερής και πολυμερής πάλι. Και εκεί ενισχύσαμε τις προσπάθειές μας ε, για διάλογο και εταιρικέ σχέσεις με χώρες που εφαρμόζουν τέτοιου περιορισμούς αλλά και που επηρεάζονται από περιορισμούς στο εμπόριο τέτοιων πρώτων υλών. Πρόκειται για έναν το κλάδο και στα πλαίσια του ΟΣΑ συνεργαζόμαστε με πολλές χώρες, μέλη του ΟΣΑ, αλλά και μη μέλη του ΟΣΑ, που συμμετέχουν σε, ένα, σε μια ομάδα εργασίας για την πρόσβαση στις πρώτες ύλες. Το σχέδιο δράσης μας στηρίζεται σε αυτούς τους τρεις πυλώνες που σας προανέφερα και τις αναλύει πιο διεξοδικά. Έχουμε ένα δεκασέλιδο έγγραφο Μερικές προτάσεις μας είναι πιο συστημικές, αναλυτικές και άλλες καλύπτουν συγκεκριμένες δράσεις. Αν θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες, ε, μπορείτε να υποβάλλετε ερωτήσεις. Τέλος, όπως θα διαπιστώσατε, οι δράσεις μας είναι πολύ σχηδείς. Εξού και η δυσκολία της εφαρμογής τους. Μερικές είναι εύκολες εφαρμογής και άλλες ε, πολύ δύσκολες. Γι' αυτό και προβλέπουμε τακτική ενημέρωση για την ε, πρόοδο και μία ετήσια έκθεση που θα εκδοθεί στα τέλη του έτους. Αυτά προς το παρόν κύριε Πρόεδρε και περιμένω τις ε, ερωτήσεις αν υπάρχουν ενδεχομένω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πολύ ενδιαφέρουσε οι παρατηρήσει σα και η εισαγωγή σα. Το έγγραφο το ίδιο είναι πραγματικά συναρπαστικό κείμενο. Καλωσορίζω θερμότατα την πρότασή σας να είμαστε σε διαρκή επαφή και συνεννόηση για αυτό το θέμα, γιατί πραγματικά ο ανεφοδιασμός και το εμπόριο σε πρώτες ύλες για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπαρξιακή σημασία. Χρειάζεται λοιπόν συνεχής ανασχόληση και παρακολούθηση του θέματος. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα κοιτάω γύρω μου. Οι συνάδελφοί μου έχουν ερωτήσεις. Είστε ικανοποιημένοι με τις ε, παρατηρήσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις εξηγήσει. Σας καλύπτουν πλήρως και συμφωνείτε απόλυτα. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Ε, και περνούμε στο σημείο 6 της της διάταξης. Όργανο ελέγχου εμπορικών πολιτικών του ΠΟΕ σχετικά με την εμπορική πολιτική των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Έχετε λάβει όλοι στα έγγραφά σας την αντίστοιχη ενημέρωση και τεκμηρίωση που έχει υποβληθεί εκ των προτέρων. Θα γνωρίζετε ότι έχει εκπονήσει η γραμματεία του ΠΟΕ ένα έγγραφο για την αναθεώρηση των εμπορικών πολιτικών. 6 με 8 Απριλίου έγινε αυτό. Και βέβαια ο έλεγχος και η παρακολούθηση από την κάθε χώρα ως προς το εμπόριο είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί θεωρούμε και γνωρίζουμε ότι η εμπορική πολιτική είναι πλέον κοινή εμπορική πολιτική αλλά στην εκτέλεσή της είναι αρμόδια τα κράτη-μέλη, έτσι. Οπότε είναι και ε, καθήκον του ΠΟΕ να ελέγχει και να παρακολουθεί με ποιο τρόπο εκτελούν και υλοποιούν τα κράτη-μέλη τα αποφασιστέντα. Κανονικά εκπονούνται δύο έγγραφα Πρώτο έγγραφο είναι τα παρακολουθούμενα εντό εισαγωγικών κράτη που δίνουν αυτές τις δηλώσεις πολιτικής ε, και ελέγχονται και μετά η ανεξάρτητη γραμματεία του ΠΟΕ δίνει το δικό της έγγραφο και, ε, μπορούμε να κάνουμε δύο σημαντικές ε, παρατηρήσεις τώρα. Το έγγραφο αυτό τεκμηριώνει και αναγνωρίζει πάρα πολύ αυτό που έχει ε, πει ανέκαθεν και η Επιτροπή Εμπορίου, ότι το πολυμερές ε, σύστημα εμπορίου είναι πραγματικά οι ρίζες για η πηγή της συνοχής μιας κοινή εμπορικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση που να έχει και συνοχή. Και προφανώ. Και θα πρέπει να προωθηθούν λοιπόν οι διαπραγματεύσεις, οι συνεννοήσεις. Ανεξάρτητα όμως από αυτά όλα θα πρέπει να διαπιστώσουμε ότι η ευρωπαϊκή κοινότητα και τα κράτη-μέλη έχουν τελείως διαφορετικό δίκτυο δυνατοτήτων και προτιμησιακών συμφωνιών που τις αξιοποιούν κιόλας. Και με τις αναπτυσσόμενες χώρες και με τις ανεπτυγμένες. Και θα πρέπει πηγόντως η γραμματεία του ΠΟΕ να το προσέξει αυτό και να μην ε, προκύπτουν από τις καταστάσεις αυτές παραβιάσεις των κανόνων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου. Ένα δεύτερο που μπορούμε να πούμε είναι το εξής γνωρίζετε ότι είναι παγκόσμιος ηγέτης, ε, εξαγωγέας δηλαδή η Ένωση σε αυτά τα θέματα και, δε, και δεύτερος εισαγωγέας παγκοσμίω. Και δραματίζουμε πολύ σημαντικό ρόλο για την οικονομική ανάπτυξη και την ανάπτυξη γενικότερα και τις ανταλλαγές και τις συναλλαγές. Και τελικά καταλήγουν ότι ενδεχομένω να υπήρχε και περαιτέρω δυνατότητα για τη γεωργική παραγωγή να απελευθερωθεί ακόμα περισσότερο, να προστεθούν οι διαδικασίες συντελωνιακές και να μειωθούν ενδεχομένω και ανώτατοι δεσμοί. Αυτό το θέμα είναι επίμαχο, επανειλημμένα. Το έχουμε συζητήσει τι κάνουμε στη Γεωργία. Στο ιστορικό του ΠΟΕ έχει γίνει μεγάλη φασαρία ότι έχουμε πολύ μεγάλες επιδοτήσεις εξαγωγικές στα γεωργικά προϊόντα, όπως κάνουν και για το βαμβάκι ας πούμε είπα και οι χώρες της Δυτικής Αφρικής που επίσης παράγουν ε, βαμβάκι ανθίστανται και ε, ήταν δυσαρεστημένοι που αρχίζουμε μόνο από το 2013 να μειώνουμε τις εξαγωγικές. Είναι πολύ επίμαχο αυτό το θέμα ακόμα στον ΠΟΕ. Γι' αυτό χαιρόμαστε πάρα πολύ που έχουμε εδώ πει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κοιτάξω λίγο στο χαρτάκι μου να σας πω και ποιο είναι. Να μας κάνει μία παρουσίαση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρώτα και μετά συζήτηση. Είναι ο κύριος Παόλο Γκαρτσότη ή η κυρία Μαρτίνα Ντράντ. Δεν ξέρω πώς θα το μοιράσετε και ποιος θα μιλήσει πρώτος. Παρακαλώ. Έχετε το λόγο. Thank you, Mr. Ευχαριστώ. Όπως βλέπετε είμαι ο κύριος Γκατζότη, όχι η κυρία που αναφέρατε. Όπως είπατε σωστά, αυτό είναι πολύ σημαντικό για την Παγκόσμια Οργάνωση Εμπορίου και για την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί ε, ο μηχανισμός αυτός εμπορικής πολιτικής είχε δυσπιστεί πριν ακόμη και το γύρο της Ουρουγουάης. Εφαρμόστηκε από το ΓΚΑΤ το 1988 μετά τη συνδιάσκεψη του Μόντρεαλ και θεσμοθετήθηκε στη Συμφωνία της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εμπορίου. Είναι πολύ σημαντικός αυτός ο μηχανισμός για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ισχύει και για την Ιαπωνία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και γίνεται αυτή, αυτός ο έλεγχος κάθε δεύτερη χρονιά. γίνεται πρώτα με την Ιαπωνία, τι Ηνωμένε Πολιτείε και την Ιαπωνία και μετά έχουμε τα 16 άλλα μέλη τη Παγκόσμια Οργάνωσης Εμπορίου κάθε 4 χρόνια γιατί δεν έχουμε τόσο σημαντικές εμπορικές συναλλαγές ε, και 6 χρόνια με τι υπόλοιπε χώρε που έχουμε ακόμη λιγότερε συναλλαγές. Καταρχήν, η γραμματεία της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εμπορίου δεν χρησιμοποιεί αυτό το, το εγχείρημα για να διαπιστώσει αν οι κοινωτικέ πολιτικές ε, συμμορφώνονται με τις διατάξεις Παγκόσμιας Οργάνωσης Εμπορίου. Αναφέρεται ότι ο μηχανισμός αυτός δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τέτοιους σκοπούς. Είναι κάτι που βρίσκεται μεταξύ των διαπραγματεύσεων και των ε, διακανονισμών διαφορών στην Παγκόσμια Οργάνωση Εμπορίου. Και ο Πασκάλα Μία, Γενικός Διευθυντής της ΠΟΕ, μιλάει για μια ενδιάμεση φάση που χαρακτηρίζεται από διαφάνεια, από ανταλλαγή πληροφοριών, πίεση μεταξύ ομοτήμων, παρακολούθηση και σε μερικέ ε, περιπτώσει είναι πολύ σημαντικό αυτό ο μηχανισμό, περισσότερο και από τι διαπραγματεύσει μερικέ φορέ και από τη διευθέτηση των διαφορών. Θα ήθελα καταρχήν να σα πω δύο λόγια για το τι συνέβη στη Γενέβη, Πώ ετοιμάσαμε αυτό το μηχανισμό και τι γίνεται με την έκθεση, ποιο είναι το περιεχόμενό της. Ήταν η ένατη φορά που η εμπορική πολιτική της Ένωσης πέρασε από αυτό το μηχανισμό επιθεώρησης. Ε, ήταν αθρώη προσέλευση στη συνάντηση αυτή, άνευ προηγουμένου, και Είχαμε λάβει πριν την ε, διάσκεψη πάνω από χίλιες ερωτήσεις για την εμπορική μας πολιτική και μάλιστα καταφέραμε να απαντήσουμε σε όλες εγκαίρως ε, και διεξοδικά. Κάτι που δεν ισχύει για όλα τα μέλη της ΠΟΕ. Η συνάντηση αυτή έγινε στις αρχές Απριλίου, 6 έως 8 Απριλίου και ο πρέσβης που προέδρευσε ήταν ο Αυστραλός πρέσβης και μάλιστα η στάση του ήταν πολύ επικοδομητική. Αναφέρθηκαν και κάποια σημεία της Γεωργίας. Κάτι που επαναλήφθηκε πάντως συζητήσει είναι ότι η διαδικασία λήψη αποφάσεων μερικές φορές εμποδίζει την, μια σωστή πρόσβαση στην ε, κοινοτική αγορά. και στα πλαίσια της χρηματοπιστωτικής κρίσης χρειάζεται μια πιο αποτελεσματική αντίδραση. Σε ό,τι αφορά τα σχόλια των μελών της ΠΟΕ και η DDA αλλά και ο, ρόλος, ο δραστήριος ρόλος της Επιτροπής της DDA ήταν πολύ σημαντικά στοιχεία. Όλοι αναγνώρισαν το θετικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εκεί. Και φυσικά ενθαρρύνθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, διαδραματίσει ηγετικό ρόλο, ιδιαίτερα στην εφαρμογή της πειθαρχία ε, δεδομένης και της κρίσης. Βέβαια, το εμπόριο δεν είναι η αιτία της κρίσης, αλλά μάλλον το θύμα αυτής της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης. Υπήρξε μια κατακόρυφη πτώση του εμπορίου. Ήδη από πέρυσι στα τέλη του έτους και για φέτος ε, ο ΠΟ υπολογίζει μείωση κατά 9% στο παγκόσμιο εμπόριο η όσα, όσα ανήγγειλε επίσημα ότι ε, οι προβλέψεις του είναι ακόμη πιο απεσιόδοξες για το 2009, 13 με 14% μείωση στο παγκόσμιο εμπόριο. Οπότε μιλούμε για δραματική πτώση στις εμπορικές συναλλαγές. Γι' αυτό είναι σημαντικό στη φάση αυτή να κρατήσουμε ανοιχτέ τις αγορές και να μην θεσπίσουμε μέτρα που να ε, παρακολύουν ε, την πρόσβαση στις αγορές ή να ενθαρρύνουν τον προστατευτισμό. Γιατί με την κρίση να σοβεί τέτοιες πιέσεις θα είναι όλο και πιο μεγάλες. Κάτι άλλο που ε, εκτίμησαν ιδιαίτερα τα μέλη της ΠΟΕ στην συνεδρίαση είναι ο ρόλος που διαδραματίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά την παραγωγή τεχνικής αλλογής και σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στην αγορά της για τις αναπτυσσόμενες χώρες, για τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες ιδιαίτερα. Και έχουμε για τις λιγότερο αναπτυγμένες οικονομίες ένα φορολόγιο το καθεστώς και προνομιακό. Και εκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κρατημέλη προσφέρουν στο πλαίσιο του προγράμματο Aid for Trade, πολύ σημαντική βοήθεια σε αναπτυσσόμενε χώρες. Είχαμε από τη Βραζιλία, Καναδά, Ινδία και Αυστραλία, τους είναι υπόπτου δηλαδή πολλά σχόλια και επικρίσεις, ενώ οι Ηνωμένε Πολιτείε ήταν πολύ πιο επίοικοι στις κριτικές τους. Είναι αλήθεια ότι η Γεωργία βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων και Σίγουρα δεν χάρηκαν όλοι με την επανεισαγωγή των εξαγωγικών επιδοτήσεων για τα καλακτοκομικά προϊόντα, δεδομένης και της κρίσης και της δέσμευσης των G20 να μην ενισχύσουν ε, πιθανά προστατευτικά μέτρα. Βέβαια υπάρχουν ε, όλο και μεγαλύτερες ανησυχίες για το ρυθμιστικό μας καθεστώς που αφορά τα βιομηχανικά προϊόντα, τις, τους τεχνικούς φραγμούς στο εμπόριο και ιδιαίτερα για τα φυτογειονομικά προϊόντα. Ιδιαίτερα ε, για τον κανονισμό REACH. Ασκήθηκαν αδρυμήτατες επικρίσεις από ορισμένου εξαγωγής για τα σημεία αυτά. Η αναθεώρηση της εμπορικής πολιτικής φυσικά είναι μια πολύ δραστηριότητα. Γίνονται πολλές συνεδριάσεις όπου όλα τα μέλη μπορούν να υποβάλουν ερωτήσεις και να λαμβάνουν το λόγο. Αλλά έχουμε και την έκθεση της γραμματείας. Η έκθεση της γραμματείας είναι μια μερόληπτη, ουδέτερη και διεξοδική ανάλυση της εμπορικής πολιτικής του μέλους του, της ΠΟΕ που ελέγχεται. Βέβαια, έχουμε δει πολύ καλύτερες εκθέσεις, πολύ πιο ποιοτικές και πολύ πιο ουδέτερες από αυτή που εκπώνησε η γραμματεία της ΠΟΕ την τελευταία φορά. Τέσσερα είναι κυρίως τα θέματα που διακρίνονται στην έκθεση της γραμματείας της ΠΟΕ. Η έκθεση βέβαια δεν υποβάλλεται άπαξ, ακολουθεί διάφορα στάδια και εξετάστηκε για ένα περίπου εξάμεινο πριν τη δημοσίευση του της, τη, Δευτέρα Μαρτίου, τη με την γραμματεία της ΠΟΕ. Έγινε ανάλυση για τη γεωργική πολιτική και δόθηκε έμφαση στα προστατευτικά μέτρα και στις εξαγωγικές επιδοτήσεις. Ήταν παραπλανητικά τα σχόλια σε σχέση με την έκθεση του 2007. Στην έκθεση του 2007 Αυστρία, για παράδειγμα, υποβλήθηκαν κάποια μέτρα που συνεχίζουν να εφαρμόζονται και πολύ σημαντική κλάδοι της γεωργίας υπέστησαν μεταρρυθμίσεις. Αυτό δεν αναφέρθηκε δεόντως στην τελευταία έκθεση της γραμματείας της ΠΟΕ. Σε ό,τι αφορά τη μεταποιητική βιομηχανία, η έκθεση την ε, θεωρεί ως σημαντικό δικαιούχο κρατικών ενισχύσεων με πολλά προστατευτικά μέτρα. Και πάλι εδώ δεν δίνεται ιδέουσα έμφαση στις τελευταίες εξελίξεις. Γιατί σίγουρα ο προστατευτισμός ε, που επιφυλάσσουμε εμείς στην ε, μεταπητική μας βιομηχανία δεν είναι ο μεγαλύτερος που παρατηρείται σε μέλη της ΠΟΕ. Οπότε οι περισσότερες παρατηρήσεις της γραμματείας της ΠΟΕ δεν είναι και πολύ αμερόληπτες ε, είναι αρκετά αιτιολογημένες γιατί δεν συνοδεύονται από παραδείγματα. Για την εσωτερική αγορά μιλούν για ένα τελές πρόγραμμα και δεν μας ικανοποιεί αυτό το σχόλιο. Φυσικά ουδής δεν είναι τέλειος, αλλά θα προτιμούσαμε στην περίπτωση αυτή η γραμματεία της ΠΟΕ να εκτιμήσει τις μέχρι τώρα εξελίξεις στην εσωτερική αγορά από το να επιμείνει μόνο στην ανάγκη περαιτέρω ολοκλήρωσης και απελευθέρωση στις υπηρεσίες, στη φορολογία, στα, στις προδιαγραφές και ούτω καθεξής. Ένα άλλο θέμα που επισήμανε η Γραμματεία είναι το περιφερε... οι συμφωνίες περιφερειακού εμπορίου, περιφερειακές συμφωνίες εμπορίου. Στο παρελθόν, και εμείς αλλά και άλλα μέλη της ΠΟΕ ασχολήθηκα με το θέμα αυτό και οι τελευταίες συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου αλλά και οι πολιτικές της ανακοίνωση για την, παγκόσμια, την παγκοσμιοποιημένη Ευρώπη ή την ολοκληρωμένη Ευρώπη δεν είναι μια πολιτική που επικεντρώνεται μόνο σε κάποιες ρηχές περιφερειακές συμφωνίες. Ήταν αρκετά μακροσκελή η έκθεση της γραμματής, γι' αυτό χρειάζεται να μακρηγορήσω κι εγώ. Πάντως, το εγχείρημα ήταν πολύ σημαντικό και οι υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής μαζί με τα κράτη-μέλη συνεργάστηκαν στενά και άοκνα για πολλούς μήνες. Και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που είχαμε την ευκαιρία να σας ενημερώσουμε. Κάτι που κάνουμε ιδιαίτερος με ιδιαίτερη χαρά για την ενημέρωσή σας των δραστηριοτήτων της ΠΟΕ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μήπως κάποιος από τους συναδέλφους σας θέλει κάτι ε, να προσθέσει, όχι, οπότε αυτή είναι η τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ για τις ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις. Αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί να μην είναι κανείς ευχαριστημένος όταν ακούει κριτικές για τις οποίες θεωρεί ότι δεν είναι αιτιολογημένες. Αυτό συμβαίνει στους ευρωβουλευτές όλη την ώρα και ιδίως διότι ανήκουμε σε διαφορετικές πολιτικές ομάδες αυτή τη στιγμή παρουσιάστηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πιστεύω ότι είναι νορμάλ και είναι κανονικό δηλαδή φυσιολογικό και δεν ε, έχει τόσο άδικο αυτό το έγγραφο ε, και εάν συμπεριφερόμαστε όπως το πράττουμε ε, τότε η στήριξή σας είναι αμφίροπη ε, διότι νομίζω ότι αναφερθήκατε προηγουμένως στις περιφερειακές συμφωνίες και είπατε ότι δεν χρειάζεται εμείς να θεωρήσουμε ότι κάναμε κάτι στραβό αλλά με την ε, Global Europe Strategy εμείς δεν συμφωνούμε θεωρούμε ότι δεν επαρκεί και δεν, αξι... δεν ε, φτάνει να ανοίγουμε τις αγορές για να έχει δυνατότητες ε, ε, μεγαλύτερες για εκποίηση των προϊόντων της η οικονομία μας αλλά διότι δεν πρέπει να σκεφτόμαστε μόνο τις ε, επιχειρήσεις αλλά διότι η στρατηγική αυτή πρέπει να λάβει υπόψη της και την ε, εξέλιξη σε διάφορους τομείς και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό και έρχομαι τώρα στο σημείο 7 εμπορικές διαπραγματεύσεις με τις χώρες κοινότητας στον των ε, άνδεων. Λοιπόν, γιατί ε, ε, αποτυγχάνουμε και δεν προχωρούμε ούτε στον ΠΟΕ ούτε στις περιφερειακές αγορές είτε πρόκειται για το Μερκοσούρα, αν πρόκειται για τη Μέση Ανατολή πάντοτε προσπαθούμε να επιβάλλουμε πρωταρχικά την οικονομική μας πολιτική και όχι τις άλλες προτεραιότητες σε Εν πάση περιπτώσει θα φτάσουμε στο σημείο αυτό. Οι συνάδελφοι έχουν μήπως ερωτήσεις. Αν όχι, ευχαριστώ και πάλι και ε, κλείνω το θέμα αυτό το 6 της ημερήσιας διάταξης και ερχόμαστε τώρα στο 7. Το 7. Εμπορικές διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της κοινότητας των Άνδεων Ξέρετε όλοι ότι η οι εμπορικές διαπραγματεύσεις ήταν ένα βασικό θέμα και προσφάτως έγινε η συζήτηση για τις οκτώ ε, συμφωνίες εταιρικές σχέσεως για ε, την ε, ακτή του Ελεφαντοστρού και το Κάρι Φόρουμ και είχαμε συζητήσει την ε, κατάσταση των διαπραγματεύσεων με τις χώρες, το, ε, ε, χώρες Άζιαν. Εχθές στο Κοινοβούλιο είχαμε μία συζήτηση για την κατάσταση των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεως και της κοινότητας των Άνδρων και ε, χαιρόμαστε ε, όπως άλλωστε είπαμε και χθε, διότι ο Ενρίκε Ρομπρέτο ε, Καστίγιο γερουσιαστής της Κολομβίας από το 2002 ήταν εχθές παρόν είναι και σήμερα παρόν και θα μας απευθύνει το λόγο ξέρετε ότι έχουμε καταρτήσει και διάφορες εκθέσεις κατά πρωτοβουλία για τη τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ενώσεως με ε, τα, τις χώρες των Άνδεων και ο δεύτερος γύρος ξεκίνησε το Μάρτιο του 2009. Ξέρετε βέβαια ότι εντός του Κοινοβουλίου αυτού υπάρχουν διάφορες απόψεις γενικώ επί του θέματος σχετικά με τις συμφωνίες ελευθέρου εμπολίου ή GSP ή GE με μεγαλύτερη έμφαση διότι ξέρετε ότι στην κοινότητα των άνδεων υπάρχει δύσκολη κατάσταση διότι μεταξύ των κρατών μελών αυτής της κοινότητος υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για το πόσο πρέπει κανείς να, να απελευθερώσει το εμπόριο και ξέρετε ότι υπάρχει μια συμφωνία ελευθέρου εμπορίου μεταξύ του, της Κολομβίας και των Ηνωμένων Πολιτειών που ακόμη δεν έχει κυρωθεί από τις Ηνωμένε Πολιτείε, ιδίω αναφερόμενη στην κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στην Κολομβία ξέρετε ότι στο Κοινοβούλιο την περασμένη εβδομάδα έγινε μία σημαντική συζήτηση εάν ε, ε, προέπει κανείς να υπάρχει προτιμησιακές συμφωνίες με τα κράτη-μέλη όταν υπάρχει μία δυσμενής κατάσταση στη χώρα και πρόκειτο για το ο Τουρκμενιστάν το οποίο είχε κλείσει τις ε, πόρτες του βία όπου υπήρχε μόνο ερυθρός σταυρός δεν υπάρχουν μη κυβερνητικέ οργανώσεις δεν υπάρχει δυνατότητα τότε να εκφραστεί κανείς ελεύθερα και αν κοιτάξουμε και την κατάσταση στην Κολομβία ε, υπάρχουν ε, διάφορες πληροφορίες οι οποίες είναι πολύ ανησυχητικές σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ιδίω οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ε, και άτομα τα οποία απασχολούνται στην εξόριξη των πρώτων υλών. Ε, ξέρετε ότι η Κολομβία είναι αποκλεισμένη γιατί ε, η ε, πνευματική ιδιοκτησία δεν καλύπτεται και αυτό είναι κάτι το οποίο ε, δεν προχώρησε. Είπαμε λοιπόν ότι είμαστε ενάντια σε αυτή τη διακοπή των συζητήσεων που είναι αντίθετη προς τους πολιτικούς στόχους μας. Ε, θα πρέπει να υπάρξουν αυτές ε, οι ε, ε, ε, οι διαπραγματεύσεις διότι βασιζόμαστε στον πολιτικό διάλογο και στη συνεργασία πρέπει να υπάρχει και ένας πυλώνας εμπόριο αλλά το πώς πρέπει αυτό να ισχύσει είναι ένα αμφιλεγόμενο θέμα διότι θα πρέπει να καλωσορίσουμε και πάλι τον γερουσιαστή Ρομπρέντο Καστήλιο. Σας δίνω δίνω κατά πρώτα το λόγο για να μας πείτε ποια είναι η δικιά σας άποψη για τις ε, εμπορικές ε, αυτές συμφωνίες. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να απευθύνω τον ιδιαίτερο χαιρετισμό μου προς τον κύριο Μάρκοφ για τη φιλοξενία του και να σας ευχαριστήσω θερμά για την ευκαιρία που μας δώσατε να παραβρεθούμε στη συνεδρίασή σας. Θα ήθελα να πω ότι η δική μου γνώμη είναι ότι η μία χώρα σαν την Κολομβία δικαιούται τις καλύτερες δυνατές διπλωματικές και εμπορικές σχέσεις με τους εταίρους της. Είμαστε υπέρ αυτών των συναλλαγών, των αγοραπολισιών, αλλά και των αλλοδαπών επενδύσεων στην πατρίδα μας, στην Κολομβία. Σε γενικού όρου λοιπόν συμφωνούμε. Άλλωστε Όλοι οι άνθρωποι νομίζω πιστεύουν ότι είναι θετικές οι σχέσεις μεταξύ των χωρών. Πιστεύουμε όμως ότι οι σχέσεις αυτές ε, δεν μπορούν να έχουν οποιαδήποτε μορφή να είναι ανεφόρων. Γιατί μερικές φορές είναι κατάλληλες, αλλά μερικές φορές είναι τελείως ακατάλληλες τέτοιες σχέσεις. Για αιώνες ολόκληρους η Αμερικανική Υπήρωση, Νοτιοαμερικανική Υπήρωση ε, ήταν υποτελής της ευρωπαϊκής κορώνας. Διεκδίκησε την ανεξαρτησία της η αυτή και την διακήρυξε, γιατί νομίζω ότι κάθε λαός δικαιούται την ανεξαρτησία του. Με αυτή λοιπόν τη διευκρίνηση ε, γιατί υπάρχουν και θετικές αλλά υπάρχουν και αρνητικές σχέσεις. Ε, θα ήθελα να πω ότι στην Κολομβία έχουμε περίπου δύο δεκαετίες ε, που εφαρμόζουμε πολιτικές που θα μπορούσαμε να τις χαρακτηρίσουμε ως πολιτικές ελεύθερου εμπορίου. Κυρίως με βάση τους κανόνες της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εμπορίου. Και ο απολογισμός που κάνουμε σήμερα από τις συμφωνίες αυτές ελεύθερου εμπορίου είναι ολέθριος, είναι ιδιαίτερα αρνητικός για τους λαούς μας γιατί διαπιστώσαμε ότι τις τελευταίες αυτές ε, δύο δεκαετίες αυξήθηκε ε, η ανεργία, η φτώχεια, η εξαθλίωση, επιδεινώθηκε η ποιότητα της απασχόλησης. Για μας λοιπόν ελεύθερο εμπόριο δεν ισοδυναμεί με πρόοδο και ανάπτυξη, αλλά δυστυχώς ε, ισούται με το αντίθετο φαινόμενο. όλες αυτές οι πολιτικές ε, του ελεύθερου εμπορίου και του αφιλελευθερισμού οδήγησε σε, στην απώλεια της βιομηχανίας μας. Παρόλο που δεν είχαμε ποτέ μια ισχυρή βιομηχανία, χάσαμε και την ε, μικρή βιομηχανία που είχαμε, γιατί ήμασταν αυτάρκης και σε παραγωγή ε, τροφίμων μέχρι το 1990, ενώ φέτο εισάγουμε πάνω από 8 εκατομμύρια τόνου τροφίμων, ενώ θα μπορούσαμε κάλλιστα να παράγουμε αυτά τα τρόφιμα στην Κολομβία. Όλα αυτά είναι απλά παραδείγματα, αλλά στην Κολομβία, για παράδειγμα, επιδεινώθηκαν οι συνθήκες παραγωγής των γενώσιμων φαρμάκων, κάτι που δυσχέρανε την πρόσβαση στα φάρμακα για ένα λαό που είναι φτωχός, που πολλές φορές είσαι σε άθλιες συνθήκες. Και μάλιστα πολλές κρατικές επιχειρήσεις, αλλά και ιδιωτικές, έχασαν τον εθνικό τους χαρακτήρα. Τα τελευταία 15 χρόνια η Κολομβία έχει λάβει 100 δισεκατομμύρια δολάρια αλλοδαπές επενδύσεις, ενώ εξήγαγε ε, ε, είτε από χρέους είτε από διάφορες άλλες υποσχέσεις 160 δισεκατομμύρια δολάρια. Δηλαδή υπήρξε μια φέμαξη του, του κεφαλαίου. Και σίγουρα η εσωτερική μας ανάπτυξη δεν οφείλεται στην, στις αλλοδαπές επενδύσεις, αλλά οι δικές μας αποταμιεύσεις ενισχύουν τις άλλες τις ξένες οικονομίες. Δεν νομίζω λοιπόν ότι είναι θετικό για την Κολομβία να εμβαθύνει τις α, α, σχέσεις της ελευθέρου εμπορίου, γιατί αν ο ΠΟΕ ήταν αρνητικός για μας, ο εσύ είναι ακόμη πιο ε, αρνητική, η είναι ακόμη πιο αρνητική κατάσταση. Εμείς θεωρούμε ότι είναι πολύ αρνητικό μια χώρα σαν την Κολομβία που είναι υπέρ των διαδικασιών ολοκλήρωσης αλλά και πάλι όρους εξαρτάται ε, με ποιες χώρες γιατί μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με τη ΣΥΠΑ ή με ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση γίνονται εις βάρος των περιφερειακών διαδικασιών ολοκλήρωσης τέτοιες ε, συμφωνίες ε, ελευθέρου εμπορίου με ΗΠΑ ΕΕ και Ευρωπαϊκή Ένωση καταστρέφουν τις δυνατότητες ε, σύναψης περιφερειακών τέτοιων συμφωνιών με την Κολομβία. Έχουμε πολλούς λοιπόν οικονομικούς και πολιτικούς λόγους και επιχειρήματα που κρίνουν ότι δεν είναι θετικές αυτές οι εξελίξεις για την Κολομβία. Ακόμη ε, και για την εθνική μας κυριαρχία υπαγόμαστε σε αποφάσεις ισχυρότερων από εμά χωρών που καθοδηγούνται κυρίως από τα συμφέροντα των πολυεθνικών τους. Σίγουρα ε, δεν θα εστερνίζονται πολύ τις απόψεις μου, αλλά θα ήθελα να προσθέσω κάτι ακόμη και ελπίζω εκεί να συμφωνήσουμε. Πρόκειται για κάτι που ε, ε πολύ σωστά ε, αναφέρθηκε. το Δημοκρατικό Κόμμα των ε, Ηνωμένων Πολιτειών αρνήθηκε να επικυρώσει τη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου, όχι για οικονομικούς λόγους, αλλά για πολιτικούς λόγους και πολύ δικαιολογημένα κατά τη γνώμη. Πολύ σωστά το Δημοκρατικό Κόμμα των Ηνωμένων Πολιτειών θεωρεί ότι η κυβέρνηση της Κολοβίας η κυβέρνηση του Προέδρου Ουρίμπε δεν ε, παίρνα εξετάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν έχει καλές επιδόσεις. Έγιναν πολλά εγκλήματα κατά το συνδικαλισμό, κατά του συνδικαλιστικού κινήματος. Μένουν ατιμόρυτα τα εγκλήματα κατά, το συνδικαλιστών, κατά των ηγετών του συνδικαλιστικού κινήματος. Και ε, δυστυχώς ε, πολλοί μέτεροι της κυβέρνησης έχουν ύποπτες σχέσεις με παρα, παραστρατητικές οργανώσεις και μεροληπτικέ δράσει και αποφάσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου, κάτι που δείχνει ότι δεν υπάρχει σαφής διάκριση εξουσιών στην Κολομβία. Και μάλιστα η κυβέρνηση προσπαθεί να αναθεωρήσει για δεύτερη φορά το Σύνταγμα της Κολομβίας για να επανεκλεγεί ο πρόεδρος Ουρίμπε, γιατί όταν αρχικά ε, εξελέγει ο Ουρίμπε η η προεδρική θητεία διαρκούσε μόνο τέσσερα χρόνια. Τροποποίησε το Σύνταγμα προκειμένου να επανεκλεγεί δεύτερη φορά και τώρα μπορεί να το ξανααναθεωρήσει. Το Δημοκρατικό Κόμμα λοιπόν των Ηνωμένων Πολιτειών θεωρεί ότι η κολοβενή κυβέρνηση δεν θα πρέπει να επιβραβευθεί για τις επιδόσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα με μια τέτοια σύναψη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου. Είναι πραγματικά Κρίμα όμως να συναυθεί τέτοια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου ε, της Κολομβίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί έτσι θα δοθεί άφεση αμαρτιών στο Ουρίμπε και θα καθαγιαστεί και θα θωθεί ο Ουρίμπε χάρη σε μια τέτοια συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, ε, δεν δέχονται να επικυρώσουν τέτοια συμφωνία. Γιατί αν η Ευρωπαϊκή Ένωση υπογράψει μια τέτοια συμφωνία με την Κολομβία θα είναι σαν να αναγνωρίζει ότι η Κολομβία σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Προσοχή λοιπόν. Πιστεύω ότι στην Κολομβία δεν θα πρέπει να συναθεί καμία συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ τη κολομβιανή κυβέρνηση και οποιασδήποτε άλλη. Ευχαριστώ πολύ, Γερουσιαστά. Πρώτη ζήτησε το λόγο η Έρικα. Παρακαλώ. Έρικα Μαν, στα αγγλικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, εκτιμώ πάρα πολύ αυτά που είπατε. Όλα όσα είπατε. Και όλες οι αναφορές που κάνατε περιγράφουν ακριβώς την κατάσταση στην Κολομβία. Θα πρέπει όμως να λάβουμε υπόψη μας επίσης το εξής. Αν δούμε με ποιον τρόπο θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση να υπογράψει μια συμφωνία με την Κολομβία, ε, ίσως δεν θα πρέπει να λησμονούμε τα εξή δύο στοιχεία. Εγώ ήμουν εδώ στο Κοινοβούλιο όταν διαπραγματευτήκαμε τη συμφωνία με το Μεξικό και θυμάμαι πάρα πολύ καλά και τη συζήτηση που είχαμε και την αντιπαράθεση με τους Μεξικανούς. Δεν ήταν η ίδια ακριβώς, αλλά πολύ κοντά ε, το ύφος. Ε, πολύ επιφυλακτική θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει το δημοκρατικό έλλειμμα και τα, ε, τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όταν θα υπογράψει τη Συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση μήπως χάσει κάποια δικαιώματα. Εγώ είμαι και πρόεδρος τώρα της αντιπροσωπείας με το Μεξικό τα τελευταία 4-5 χρόνια. Ε, πιστεύω ότι παραμένουν ε, εμφιβολίες, δεν έχουν διαλυθεί και θα παραμείνουν ακόμα διότι δεν υπάρχει η απόλυτη αλήθεια. Ποιο είναι το απόλυτα σωστό, να υπογράψει κανείς ή να μην υπογράψει. Δεν υπάρχουν απόλυτα εργαλεία ε, ό,τι και να κάνει κανείς στη ζωή αναλαμβάνει κάποιο κίνδυνο. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει περισσότερα δικαιώματα παρέμβασης ακριβώς ε, μετά από την υπογραφή διότι έχουμε ρήτρα για τα ανθρωπίνα δικαιώματα διότι τη στιγμή που υπογράφουμε τη συμφωνία αναλαμβάνουμε και ευθύνη. Και εδώ έχω τις περισσότερες επικρίσεις, αν θα πρέπει να το πράξουμε. Γιατί τη στιγμή εκείνη που παίρνουμε τις ευθύνες μας, Ε, μπαίνουμε και σε κάποιες διαδικασίες και εκεί έχω πάντα κάποιες ε, επιφυλάξεις με χώρες που δεν έχουν τελείως δημοκρατικά στάνταρ και προδιαγραφές. Πρόεδρε, τι γίνεται, έχετε πρόβλημα χρόνου. Εντάξει, να συντομεύετε, δείχνει ο πρόεδρος. Ε, πάντα είναι δύσκολο να κάνουμε συζήτηση αν δεν μπορούμε να ε, ε, εξηγούμε τα θέματα. Πάντως, επειδή ε, ε, αναφερθήκατε στη δημοκρατική σκοπιά αυτή, ε, συμφωνώ απολύτως, αλλά σας αντιστρέφω το ερώτημα. Διότι δεν υπάρχει άσπρο μαύρο. Μήπως είναι καλύτερα να έχουμε συμφωνία και βάσει τη συμφωνία αυτής να προσπαθούμε να βοηθήσουμε την Κολομβία να, να αναπτύξει περισσότερες ε, δημοκρατικές προδιαγραφές και ανθρώπινα δικαιώματα ή να αρνηθούμε και να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Ο πρόεδρος. Έρικα, ξέρεις ότι λυπάμαι πάρα πολύ πάντα, αλλά αυτό το θέμα που είπες είναι διολογημένο και η ερώτηση. Ε, και σε άλλες συμφωνίες προτιμησιακές έχουμε ε, δημοκρατική ρήτρα και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ρόμπερτ, εσύ είσαι ο επόμενος, Εύανς. Στέρτη, συγγνώμη. Ε, μισή ώρα κάθομαι, αλλά θα είμαι πολύ σύντομο. Ε, εγώ θέλω να ακούσω όλου. και του πρέσβεις πριν τοποθετηθώ, όχι έναν μόνο, πριν μιλήσουν τα μέλη. Όχι πρόεδρε, θα τελειώσω. Κάθομαι εδώ μισή ώρα και ακούω τη συζήτηση και μας λέτε τώρα ότι δεν έχουμε χρόνο να μιλήσουμε. Πρόεδρε, δεν είναι δίκαιο αυτό και σωστό. Είτε θέλετε συζήτηση, είτε δεν θέλετε συζήτηση για αυτό το θέμα. Και υπό την ηγεσία του Άλβαρο Ρίμπε είδαμε τι έγιναν. Αλλά έχω την εντύπωση ότι κάνει καλή δουλειά ο άνθρωπος, δεν ξέρω, διορθώστε. Έχουν μειωθεί δολοφονίες, έχει βελτιωθεί η κατάσταση στις εκβιάσεις και ε, στις απαγωγές και από ό,τι φαίνεται η χώρα σιγά σιγά βαίνει προς ένα μεγαλύτερο εκδημοκρατισμό και από ό,τι στο παρελθόν. Και εκπλήσουμε που ακούω επιθέσεις εναντίον του κυρίου Ρίμπε. Δεν ξέρω, θέλω να ακούσω και τον πρέσβη για να έχουμε ισορροπημένη ε, προσέγγιση και παρουσίαση. Αυτό για το οποίο εγώ ανησυχώ είναι το εξή. Όπως είπε και η Έρικα, αν θέλουμε να προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε από τις χώρες αυτές, και δεν ομιλώ μόνο για την Κολομβία, υπάρχουν πολλές χώρες ε, στο ε, σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων συν GSP+, κάτι πρέπει να κάνουμε. Το λέει και η Έρικα αυτό. Ε, ανοίγουμε τις αγορές, αλλά αυτό σημαίνει και μια πειθαρχία. Δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή να αποφασίζει κάποια πράγματα και να μην γίνονται σεβαστοί οι κανόνες. Και εκπλήσωμαι που ακούω τους ομιλητές να λένε ότι δεν θέλουν. Για το πετρέλαιο και για άλλα προϊόντα θα πρέπει να το κοιτάξουμε να ακούμε το σύνολο της ιστορίας, όχι μονόπλευρα ε, επιχειρήματα. Ευχαριστώ. Ρόμπερτ, θα σου απαντήσω αμέσως και βέβαια θα μιλήσει ο πρέσβης Κολομβίας, αλίμονο. Απλώς νόμιζα ότι θα ήταν πιο πρόσφορο να κάνουν ε, οι βουλευτές πρώτα τα σχόλιά του για να μπορέσει να απαντήσει ο πρέσβης και να τοποθετηθεί. Δεν έχει καμία σχέση αυτό με αδικία. Λοιπόν, δεν προσπάθησα να υποβαθμίσω κανέναν, προσπάθησα να είμαι πάντοτε δίκαιος, καλέσαμε κάποιον ο οποίος μίλησε, μετά μιλάν, μιλούν οι ευρωβουλευτές, μετά ο πρέσβης και μετά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή, πολύ σημαντικός ο προβληματισμός αυτός ο οποίος προτείνεται διότι προτείνω παρά όλα αυτά ότι πολιτιστική και ε, Οικονομική Επιτροπή έτσι όπως παρουσιάστηκε από τον γερουσιαστή δεν παρουσιάζεται σωστά διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διαπραγματεύεται με πολλές χώρες ανά τον κόσμο, χρησιμοποιεί διάφορες μεθόδους, βρίσκει διαφορετικές λύσεις είτε πρόκειται για την προσπάθεια καταρτήσεως μίας πολυμορφίας είτε αν πρόκειται ε, για μία διμερή αντιμετώπιση. Ε, τα δικαιώματα του ανθρώπου δεν είναι μία επιπρόσθετη προσπάθεια αλλά με αυτόν τον τρόπο η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να συνδιαλλαγεί με τον κόσμο και να εξάγει ανά τον κόσμο. Άρα αυτά που ζητούμε από την Κολομβία δεν πρέπει να είναι διαφορετικά από αυτά που ζητούμε από τους υπολείπους. Και θέλω να υπενθυμίσω την, ε, ε, εξαφάνιση των ε, χριστιανών στην Ινδία, αλλά κανένας δεν θα αφισβήσει συζητήσει ότι η Ινδία είναι δημοκρατική χώρα παρόλο που έχουν ε, εκριζωθεί οι ε, χριστιανοί και αυτό δεν μπόρεσε να γίνει χωρίς ε, τη συμπεγνία των αρχών. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε υιοθετήσει πολύ σημαντικές συμφωνίες με τις χώρες της Αφρικής όπου υπάρχει υπάρχει πρόβλημα με τις κυβερνήσεις. Αυτό βέβαια δεν δικαιολογεί αυτό που γίνεται στην Κολομβία το οποίο είναι κατακριτέο και πρέπει ε, η κατάσταση αυτή να παρακολουθείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Κολομβία όπως και σε όλες τις χώρες που υπογράφονται συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών και εταιρικής σχέσεως δεν λαμβάνει υπόψη της της, ε, της που έχουν επιτευχθεί διότι με αυτόν τον τρόπο μειώθηκαν σημαντικά οι ε, δολοφονίες και η ατιμορρησία. Τα δικαστήρια ε, λειτουργούν καλύτερα, έχουν γίνει πιο αντικειμενικά και ξέρουμε ότι ο αγώνας για να καταρτιστεί ένας, μια πλήρης δημοκρατία ίσως δεν επιτυγχάνει κάνετε όπως εμείς το θεωρούμε στην Ευρώπη και η Κολομβία βγαίνει από μια πολύ περίπλοκη κατάσταση και δεν μπορούμε να σκεφτούμε ότι όλες οι χώρες θα μπορέσουν να λύσουν όλα τα προβλήματα από τη μια μέρα στην άλλη διότι τότε θα μπορούσαμε να συζητήσουμε ε, τα δικαιώματα του ανθρώπου στη Βρασιλία όπου υπάρχει εξαφάνιση των ηθαγενών πληθυσμών ε, με την ε, συμμετοχή της κυβέρνησης κυβερνήσεως για να υπάρξει αποψήλωση των δασών. Λοιπόν, ε, ή χρησιμοποιούμε δύο μέτρα και δύο σταθμά ή χρησιμοποιούμε ένα κριτήριο και ζητούμε από τις χώρες αυτές να παρακολουθούνται οι ρήτρε αυτές και να διακόπτουμε την εφαρμογή των συμφωνιών εάν τα στοιχεία αυτά δεν γίνονται σεβαστά και το λέγω διότι είμαι κάποιος ο οποίος θεωρεί ότι είναι στην αντιπολίτευση σε σχέση με τις αρχές της Κολομβίας αλλά βλέπω τι συμβαίνει με τα ανθρώπινα δικαιώματα και στον υπόλοιπο κόσμο Υπάρχουν περίπου 200 κράτη ε, στον κόσμο και εκ των οποίων κάπου 50 δεν σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Συμφωνώ λοιπόν με την Έρικα Μαν ότι πρέπει να είμαστε ε, πολύ αυστηροί σχετικά με την εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά τότε δεν θα μπορούσαμε να ε, έχουμε αυτές τις συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου και που επέτρεψαν σε περιθωριακές χώρες να έχουν προσβάσεις σε διεθνείς αγορές και δεν μπορούμε να δεχθούμε αυτή τη λογική για το μέλλον τίνοντας συμπληρωματικούς κανόνες. Θα πρέπει λοιπόν οι κανόνες αυτοί να ισχύσουν. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα ο πρέσβης της ε, Κολομβίας. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να απευθύνω ε, πολύ εγκάρδιο χαιρετισμό προς τους ευρωβελευτές και στον Στυριστή Ροβλέδο και να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δίνετε να τοποθετηθώ σύντομα ως πρέσβης της Κολομβίας επί του θέματος που σας απασχολεί. Όπως γνωρίζουν όλοι, εδώ και χρόνια η Κολομβία πλήττεται από μία βία που ε, μας πονάει όλους εμάς τους Κολομβιανούς. Αυτή η βία σε μεγάλο βαθμό οφείλεται σε ένοπλες παράνομες ομάδες που χρηματοδοτούνται από το λαθρεμπόριο των ναρκωτικών, από απαγωγές και εκβιασμούς. Μετά από τη βία αυτή που εμείς οι Κολομβιανοί εμείς ε, απορρίπτουμε, πρέπει να σας πω ότι εδώ επλήγησαν οι πάντες. Πολιτικοί ηγέτες, δάσκαλοι, συνδικαλιστές, ιερείς, ε, επιχειρηματίες, ε, τοπικοί πολιτικοί ε, κυβερνήτες ήταν θύματα. Δηλαδή έθιξε όλους τους τομείς της κολομβιανής κοινωνίας η βία αυτή, δυστυχώς. Και δεν πλήττει μόνο ένα, δύο, τρεις συγκεκριμένους τομείς της κοινωνίας μας. Για να βελτιωθεί λοιπόν η κατάσταση αυτή, η ε, κολομβιανή κυβέρνηση που γνωρίζει την υποστήριξη της ε, συντριπτικής πλειοψηφίας των Κολομβιανών και τονίζω, αγαπητοί Ευρωβουλευτές, συντριπτική πλειοψηφία των Κολομβιανών υποστηρίζει την κυβέρνηση. Ε, έθεσε σε λειτουργία την πολιτική ευθύνη δημοκρατισμού με αποτελέσματα και αναγνώριση και ευχαριστώ στους μέρους που τα είπαν αυτά εξ ονόματος και της Κολομβίας και της κολομβιανής κυβέρνησης. Αυτές οι βελτιώσεις είναι προφανείς. Υπάρχουν στοιχεία για να το υποστηρίξουν. Μπορούν να αναλυθούν, να μελετηθούν. Βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο. Προχωρούμε. Βεβαίως και απομένουν πολλά ακόμα να γίνουν. Εδώ έγινε λόγο προηγουμένω, το γεγονό ότι η Κολομβία δεν περνάει, κόβεται στα ανθρώπινα δικαιώματα στι εξετάσει. Είναι καλό να θυμίσει κανεί ότι η διεθνή κοινότητα στην οποία ανήκουν όλα τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση και προφανώ και βεβαίω η Κολομβία έχουν ένα μηχανισμό που έχουν συμφωνήσει για να γίνονται αυτέ οι εξετάσει για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και ποιο είναι αυτό το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών και μέσω μια διαδικασία που ονομάζεται ε, παγκόσμια περιοδική εξέταση. Ε, έχει νόημα να πούμε εδώ ότι η Κολομβία πρόσφατα ως υπεύθυνο μέλος που είναι της διεθνούς κοινότητας έκανε, πέρασε αυτή την εξέταση ε, στην αρμόδια επιτροπή. Άκουσε πάρα πολλές χώρες να τοποθετούνται. Έδωσε τις απαντήσεις και τις εξηγήσεις. ανέλαβε τις υποχρεώσεις εκείνες που θεωρούνται απαραίτητες και μετά την εξέταση αυτή από τη ε, διεθνή κοινότητα πέρασε τις εξετάσεις αυτές η Κολομβία. Ικανοποιητική ήταν η έκφαση. Ξέρουμε βέβαια πάντα ότι μπορούμε και πρέπει να κάνουμε μεγαλύτερες προσπάθειες και θα το πράξουμε κιόλας. Και είναι καλό να γνωρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ ότι υπάρχει μεγάλη ανησυχία για τα ανθρώπινα δικαιώματα και συμφωνούμε. Πρόσφατα, μετά από την πρωτοβουλία της Κολομβίας, που συνέπεσε και με μια απόφαση που έλαβε η Ευρωπαϊκή Ένωση τέθηκε σε ισχύ ένας διάλογος διμερής Ευρωπαϊκής Ένωσης Κολομβίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Με ε, πολύ μεγάλη μερίσια διάταξη ανοιχτή για διμερή εξέταση, διμερή ανάλυση όλων των ε, καταστάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και από πλευρά Ένωση και από πλευρά Κολομβία. Συμπέρασμα και συνοπτικά. Η Κολομβία σέβεται όλου του μηχανισμού εδώ τη διεθνού κοινότητα. Υπόκειται και υποβάλλει τον εαυτό τη στον έλεγχο και στην ανάλυση. Έχει δώσει και διμερεί απαντήσει και έχει αναλάβει και την πρωτοβουλία. Όπω πρόσφατα φάνηκε, υιοθέτησε νέου μηχανισμού προ την κατεύθυνση αυτή. Τώρα, για το εμπόριο, θέλω να είμαι πάρα πολύ σύντομο, διότι γνωρίζω ότι δεν υπάρχει πολύς χρόνος. Ήρθε και η κυρία Άστον και τη χαιρετώ εγκάρδια κι εγώ. Η Κολομβία θέλει να οικοδομήσει κανόνες, σταθερούς κανόνες για την ανάπτυξη των σχέσεών της στο μέλλον με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό μας ενδιαφέρει η εμπορική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κολομβιανή κυβέρνηση, επαναλαμβάνω, υποστηρίζεται από την συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών και πιστεύει στις αρετές του ελευθέρου εμπορίου και στα δίκτυα για την προστασία των επενδύσεων και του εμπορίου. Πιστεύει στην ανάγκη να έχουμε συμφωνίες για να αποφύγουμε τη διπλή φορολόγηση για το εμπόριο, ε, αν διευρυθεί, αν διευρυθούν οι επενδύσεις, δημιουργία θέσεων απασχόλησης, ε, δημιουργία επιχειρήσεων. Ε, χρειάζεται για να ξεπεραστεί η φτώχεια και να εδρεωθεί ε, η θεσμική οικοδόμηση της χώρας. Σε ό,τι αφορά τώρα την Επιτροπή, θα πρέπει να ξέρουμε ότι η ελαστικοποίηση του συστήματος που καλά έκανε και δέχτηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση από τη μια δεν είναι επιβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι απάντηση σε διάφορα ε, ζητήματα που έθεσαν οι χώρε των Άνδεων. Μεταξύ αυτών είναι και η Κολομβία, διότι είχε οδηγηθεί σε παράλυση η διαπραγμάτευση με το σχήμα μπλοκ από μπλοκ σε μπλοκ, δηλαδή οι κρατών. Είπαμε να ελαστικοποιηθεί η κατάσταση. χώρε που θέλουν να προχωρήσουν να το κάνουν, χωρίς να αποκλειστεί κανένας από τη κοινότητα των άνδεων. Ε, ολοκληρώνω. Είναι καλό να γνωρίζουμε ότι υπάρχει νέα δυναμική με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών και θα συνεχίσουμε ε, τις διαπραγματεύσεις με τις διάφορες ε, χώρες του κόσμου για να συνεισφέρουμε προς την κατεύθυνση αυτή πραγματικά να είναι το εμπόριο πιο αποτελεσματικό, πιο ενεργό με περισσότερες επενδύσεις και περισσότερες ε, θέσεις απασχόλησης. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δώσετε να σας μιλήσω, Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρέσβη. Προτείνω την εξής διαδικασία τώρα. Δεν θα καλέσω τώρα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διότι ήρθε η Επίτροπος και η Επίτροπος θα έπρεπε να μας πει ε, ποιες, ε, ποια είναι η κατάσταση των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεως και Κοινότητας των Άνδεων και ε, βλέπετε υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Πάντοτε υπήρχαν, πάντοτε θα υπάρχουν. Υπάρχουν στην Κολομβία, υπάρχουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υπάρχουν μεταξύ των ε, εκπροσώπων των μη κυβερνητικών οργανώσεων και των ε, ευρωβουλευτών είναι δημοκρατικό και σωστό. Ευτυχώς μπορούμε να συζητήσουμε έτσι μεταξύ μας. Πρέπει να συζητούμε έτσι και είναι κατανοητό ότι η αξιολόγηση ε, των, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι κάτι το οποίο πρέπει να συζητείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι ο κατάλληλος χώρος ε, και μπορούμε να συζητήσουμε διάφορα θέματα εδώ και έχουμε και την ρήτρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων την οποία μπορούμε να αξιολογήσουμε. Ε, ευχαριστώ λοιπόν όλους για τη συζήτηση. Τώρα θα εγκαταλείψω αυτό το θέμα της ημερήσιας διάταξης και θα έρθω στο 8 την κατάσταση των ενεξελίξη διεθνών εμπορικών διαπραγματεύσεων. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω την ε, Επίτροπο διότι στην τελευταία συνεδρίασή μας ήρθε, δηλαδή σήμερα, για να μας παρουσιάσει τις ε, πιο ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των εμπορικών διαπραγματεύσεων και την ευχαριστώ για την πολύ καλή συνεργασία μαζί της και την Επίτροπο και όλη την ε, και όλους τους συνεργάτες της. Ε, ευχαριστώ. Ε, μου είχατε υποσχεθεί στην πρώτη ακρόαση όταν ήμασταν σκεπτικοί ορισμένοι από εμά για το τι θα γίνει με την νέα επίτροπο και τότε ε, αυτά τα οποία υποσχεθήκατε τα τηρήσατε. Μας είπατε ότι θα έρχεστε συχνά εδώ, θα συζητάμε τα θέματά μας. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτά και σας δίνω μέσω το λόγο. Καταρχήν, θα ήθελα να σας πω ότι αισθάνομαι ε, ε, λυπούμε ότι σας χαιρετώ σαν πρόεδρο της Επιτροπής γιατί νομίζω ότι από τους ευρωβουλευτές είσαστε ο μόνος ο οποίος σίγουρα δεν θα επανέλθει θα δούμε τι θα γίνει με τις εκλογές ε, ξεκινώ λοιπόν και θέλω να σας πω ότι όταν ήρθα εδώ θυμάμαι ότι είχα χτυπήσει την πόρτα σας και εσείς μου είχατε παρουσιάσει τα διάφορα θέματα που ενδιαφέρουν την Επιτροπή και αυτό με βοήθησε να, παρουσι... να προετοιμάσω την ακρόαση. Θα μου λείψετε πολύ λοιπόν. Δεν ξέρω εάν θα επιστρέψετε στις εκλογές. Ελπίζω αν όχι να έχω την ευκαιρία να σας δω είτε στη Γερμανία ή στην επόμενη σας σταδιοδρομία διότι χάρηκα πάρα πολύ για την συνεργασία που είχαμε κατά τις συζητήσεις της Επιτροπής σας. Θα ήθελα εδώ να συνοψίσω σχετικά με την κατάσταση των θεμάτων που απασχολούν αυτή την Επιτροπή. Δεν θα μπορέσω να τα καλύψω προφανώς όλα, αλλά κατά τις ερωτήσεις και απαντήσεις θα, μπορέσουμε, θα μπορέσετε ίσως να με ρωτήσετε για τα χαρτοφυλάκια τα οποία δεν θα έχω καλύψει. Μην ντραπείτε λοιπόν να με ρωτήσετε διότι θα προσπαθήσω να σας καλύψω στο δυνατόν περισσότερα θέματα. Ε, όπως είπα στην αρχή της θητείας μου και της συνεργασίας μου μαζί σας η κρίσιμη σχέση για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η προσπάθεια να ολοκληρωθεί ο γύρος της Ντόχα και αυτό συνεχίζει να είναι στο προσκήνιο των εργασιών μας. Οι αριθμοί τους οποίους είδα από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αυτή την εβδομάδα είναι ότι το Διεθνές εμπόριο από 9% τώρα μειώθηκε στο 11% και ε, αυτό, αυτοί οι αριθμοί αποτελούν δυσκολίες όχι μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά όσοι από εσά ταξιδεύουν διεθνώς αντιλαμβάνονται το ίδιο πρόβλημα υπάρχει στις υποανάπτυξη χώρες. Πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να προωθήσουμε τις πολυμερείς διαπραγματεύσεις για να ολοκληρώσουμε τον γύρο της Ντόχα. Και ε, οι προσπάθειές μου έχουν εστιαστεί εις ε, την διαμόρφωση των σχέσεών μας με την νέα κυβέρνηση στην Αμερική με τον ε, πρεσβευτή ο οποίος είναι ο νέος εμπορικός εκπρόσωπος. Είχα την ευκαιρία να τον συναντήσω και να μιλήσω μαζί του και επίσημα και άτυπα. Του ξαναμίλησα την περασμένη εβδομάδα και είναι μια βασική σχέση διότι δεν είναι μόνο ο πιο βασικός ε, εταίρος μας εμπορικά αλλά διότι οι Αμερικανοί μπορούν να συμβάλλουν στην πρόθεση του γύρου της Ντόχα και ελπίζουμε ότι τις ε, επόμενες εβδομάδες θα μπορέσει να αξιολογηθεί ότι ε, ό,τι καλό ε, υπάρχει και οφείλεται στις Ηνωμένε Πολιτείες θα προωθηθεί στη Γενέβη για να μπορέσει να ολοκληρωθεί. Βεβαίως υπάρχουν και εκλογές στην Ινδία που είναι ένα βασικό θέμα, δεν ξέρω ποια θα είναι η έκβασή τους, αλλά θα πρέπει μόλις ε, ολοκληρωθούν να ε, επισκεφθώ τον νέο Υπουργό Εμπορίου για να προσπαθήσω να τον πείσω να επανέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Είναι λοιπόν βασικά θέματα από αυτά τα οποία συζητούμε και ελπίζω ότι ο Πασκάλ Λαμή ε, θα συμμετάσχει εις ε, τις ε, ψηφοφορίες. Δεν ξέρω αν θα συνεχίσει να είναι διευθυντής του ΠΟΕ, αλλά εν πάση περιπτώσει ελπίζω ότι θα συνεχίσει. Επιπλέον έχουμε διάφορες διμερείς συζητήσεις και ε, σήμερα συζητάτε τις σχέσεις με την κοινότητα των Άνδεων πράγμα το οποίο θα μας απασχολήσει και τα επόμενα έτη. Δεν έχω ψευδεστήσεις ε, για τα προβλήματα. Έχω συναντηθεί δύο φορές με τον πρέσβη της Κολομβίας και πρέπει να δούμε πώς θα προωθήσουμε με την ενότητα των εθνών αυτών αλλά και δίμερος στα θέματα που συζητήθηκαν σήμερα εδώ και ορισμένα από αυτά είναι πολύ σημαντικά. Ε, όσον αφορά τις ε, διμερείς ε, εμπορικές συμφωνίες υπάρχει αυτή με την Νότιο Κορέα η οποία ολοκληρώνεται. Ξέρω ότι η Επιτροπή επανήλθε προσφάτως από την Κορέα. Δεν μπόρεσα ακόμη να συζητήσω μαζί τους. Ίσως όμως μπορούν να μας ενημερώνουν. Αλλά ελπίζω ότι θα μπορέσει να ολοκληρωθεί για δύο λόγους. Καταρχήν καταρχήν οικονομικά είναι μια πολύ καλή δυνητική συμφωνία για την Ευρωπαϊκή Ένωση για πάρα πολλές βιομηχανίες. Δεύτερον, διότι είναι η πρώτη ε, συμφωνία ελευθέρου εμπορίου στον 21ο αιώνα στην οποία συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, έχουμε και επιθετικά και αμυντικά συμφέροντα. Εάν λοιπόν προχωρήσουμε προχωρήσουμε σε τέτοιες διμερές συμφωνίες οι οποίες να λειτουργήσουν θετικά για ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη θα είναι ένα καλό σημείο και γι' αυτό βλέπετε ότι προχωρούμε σε διαπραγματεύσεις με τον Καναδά για διμερή συμφωνία μια συμφωνία που δεν θα είναι εύκολη διότι ε, θα έχουμε προβλήματα παραδείγματο χάρη για να συμφωνήσουμε στη Γεωργία αλλά και πάλι θα είναι ένα βασικό σημάδι διότι είναι κάτι στο οποίο ο Καναδάς αποδίδει μεγάλη σημασία και θέλουν να προωθήσουν τις προτάσεις τους και να εξασφαλίσουν ότι η ομοσπονδιακή μορφή της κυβερνήσεώς τους θα μπορέσει να επεξεργαστεί τα θετικά σημεία, δηλαδή να παρακολουθήσουν και διάφορες πολιτείες. Όσον αφορά τις χώρες ΑΣΕΑΝ προσπαθούμε να αναπτύξουμε μία προσέγγιση ώστε οι χώρες οι οποίες αυτή τη στιγμή μπορούν να αρχίσουν διαπραγματεύσεις να μπορέσουν να το πράξουν χωρίς να απομακρυνθούμε από το βασικό μας μέλημα που είναι η περιφερειακή ολοκλήρωση και για τις οικονομίες αλλά και για να διευκολυθούν οι εμπορικές σχέσεις και η, Κεντρική Αμερική όπου τα ορισμένα προβλήματα έχουν τώρα επιληθεί και έχουν ξαναρχίσει διαπραγματεύσεις και ελπίζουμε ότι θα τις ολοκληρώσουμε όσο δυνατόν πιο σύντομα. Έχουμε δε σημαντικές ε, προσμονές. Ε, μία σύντομη λοιπόν ενημέρωση για, τις, ε, όχι όλες αλλά τις περισσότερες διμερείς συνεργασίες συνεργασίες οι οποίες έχουμε. Όσον αφορά τις εταιρικές σχέσεις ε, είχα συμμετάσχει στις συζητήσεις με τις χώρες ΑΚΕ έχουμε και περαιτέρω συζητήσεις και ελπίζω ότι την άλλη εβδομάδα θα υπογραφεί η συμφωνία και ξέρω ότι ορισμένοι από εσά θα έχετε δει την εργασία που έχουμε κάνει και ε, για να διασκετάσουμε τις ανησυχίες που δεν είναι αιτιολογημένες των χωρών ΑΚΕ αλλά και για να τις καθησυχάσουμε. Και και ε, Προσφατά ε, στην Λουσάκα εν ονόματι της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε, δέσμευσα 115 εκατομμύρια ευρώ για να προωθηθεί ένα πρόγραμμα το οποίο θα διευκολύνει το εμπόριο για να ανοίξουν μένει αγορές αλλά αν δεν μπορούν να προωθήσουν τα προϊόντα τους ως εμάς δεν θα έχουν κανένα όφελος. Ήθελα λοιπόν να συζητήσω με τις χώρες αυτές τις ανησυχίες τους, να συζητήσω συζητήσω και με την Παγκόσμια Τράπεζα και ε, μισό ε, δισεκατομμύριο δολάρια δεσμεύτηκαν ε, για να προωθήσουν τις μεταφορές. Επίσης όσον αφορά τη διέλευση των συνόρων λόγω του οδικού συστήματος και των τελωνιακών σταθμών ορισμένοι καθυστερούσαν 15 μέρες. Δεν πρέπει λοιπόν απλώς να υπάρχουν εμπορικές διευκολύνσεις αλλά ε, ε, θα χρειαστεί να δοθεί βοήθεια για να ε, ξεμπλοκάρουν οι οδηγοί που έχουν παραμείνει στα σύνορα αυτά εδώ και δύο εβδομάδες. Δεν φτάνει λοιπόν απλώς να συνάπτουμε τις συμφωνίες αλλά πρέπει να τις υποστηρίζουμε για να εξασφαλίσουμε ότι οι χώρες αυτές θα μπορέσουν να εμπορευθούν επιτυχώς και ε, ιδίως στη δυσμενή οικονομική κατάσταση που αντιμετωπίζουμε τα θέματα αυτά είναι βασικά. Το τελικό θέμα που πρέπει να πω είναι ότι τόνισα ε, πόσο στηρίζουμε τις μικρές επιχειρήσεις. Όταν λοιπόν κοιτάξτε τις στατιστικές θυμάμαι ότι στην ε, προετοιμασία ε, της ακρόασης είδα ότι μόνο 8% των χωρών εμπορεύονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για τις πιο μεγάλες εταιρείες και οι μικρέ είναι αυτέ που υποφέρουν και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να προσπαθήσει ε, να στηρίξει τις μικρές επιχειρήσεις κατά τρόπον ώστε να μπορέσουν να τις βοηθήσουμε, να τους εξηγήσουμε πώς μπορούν να εμπορευθούν και να έχουμε ε, στις ε, εμπορικές συμφωνίες τις μικρές επιχειρήσεις υπογραμμισμένε για να μπορέσουν να Μία σύντομη λοιπόν παρουσίαση της εργασίας ε, η οποία με έχει απασχολήσει πρώτα αρχικά. Ξέχασα πολλά, είμαι στη διάθεσή σας να τα συζητήσω, αλλά ελπίζω ότι είδατε ποια είναι η κατεύθυνση που θα ακολουθήσει αυτή η Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Σας ευχαριστώ βεβαίως και προσωπικά για την τόσο ε, μεγάλη καλοσύνη που είχατε για τα καλά σας λόγια και τα Ανταποδίδω. Ελπίζω να κάνει ό,τι μπορεί η κυβέρνησή σα για να παρέμει βαρόνια στον Επίτροπο και στην επόμενη θητεία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διότι πιστεύω πραγματικά ότι είναι πάρα πολύ καλή η συνεργασία μα Υπήρξε τουλάχιστον θαυμάσια. Ρόμπερτ Στέρντι, ορίστε, είσαι ο πρώτο ομιλητή μα. Σα ευχαριστώ και καλώ ήρθατε κύριε Επίτροπε. Συμμερίζομαι αυτό που είπε ο πρόεδρος μας για την θέση σας. Φυσικά δεν εξαρτάται από εσά, αλλά από τον Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου για το κατά πόσο θα κρατήσετε τη θέση σας. Με το διορισμό του Πασκάλα, νομίζω σήμερα θα γίνει η ψηφοφορία, οι περισσότεροι από εμά θα ήθελαν να εξασφαλιστεί μια συνέχεια, πολλό δε μάλλον που αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλο άγχος ε, και ένταση με τους G20 και αλλού. Αν το συναντήσετε λοιπόν, παρακαλώ διαβιβάστε το σχόλιο μου και τις ευχές μας ε, για καλή επιτυχία. Σε ό,τι αφορά την κατάσταση με την Νότια Κορέα, μήπως θα μπορούσατε να με διαφωτίσετε στο σημείο αυτό για την κατάσταση σε ό,τι αφορά την απόσυρση του δεσμολογικού καθεστώτος. Σε πρόσφατη συνάντηση των βιομηχανιών θεωρήθηκε ότι αυτό το καθεστώς το ήταν σημαντικό κόλλημα και θα κοστίσει στην αυτοκινητοβιομηχανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση 150 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Ιδιαίτερα σε μια στιγμή που ε, ο κλάδος αυτός βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση οι Νοτιοκορεάτες θα συνεχίσουν με το δεσμολογικό αυτό καθεστώς ή μήπως ε, θα τους επιτρέψει η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχιστεί αυτό το καθεστώς. Υπάρχουν διαπραγματεύσεις με την Νότια Κορέα για αυτό το θέμα. Ε, δεν ξέρω αν θα προλάβετε να έχετε καλοκαιρινές διακοπές φέτος. Θα συνεχιστούν ε, εντατικά οι διαπραγματεύσεις στο γύρο της Δόχα το, το επόμενο εξάμεινο γιατί φαντάζομαι ήδη είχατε προπαρασκευαστικέ ε, συναντήσει. Πιστεύετε ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι έτοιμε και πρόθυμε για μια συμφωνία με, για τη διεκπαιρέωση του κύριου τη Ντόχα. Ποια είναι η προσωπική σα εκτίμηση, Α, αν ήταν κατεφατική απάντηση, εμείς θα την παρθέσουμε την Επίτροπο, δεν υπάρχει πρόβλημα. Η Έρικα, επόμενη, παρακαλώ. Um, Κυρία Επίτροπε, χαίρομαι ιδιαίτερα ε, που ήρθατε στη συνεδρίασή μας και η προσωπική μου ευχή είναι να σας ξαναδούμε. Και αν μπορούμε να ασκήσουμε την πυθό μας στις συμπατριώτες για να πολύ ευχαρίστως. Ελπίζω να είναι αίσια η έκβαση του γύρου της Ντόχα. Είμαστε στο πλευρό σας πάντως, αλλά τα πράγματα δεν είναι και πολύ ελπιδοφόρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί στη Washington όλοι μπορεί να λένε καλό θα ήταν να διεκπαιρεωθεί ο γύρος, αλλά δεν ξέρουμε με ποιο τρόπο. Δεν έχει οριμάσει ακόμη η κατάσταση. Θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που θα πρέπει να συναντηθεί με ομολόγους του στο Κογκρέσο, γιατί εκεί υπάρχουν ε, επιφυλάξεις. Και κυρίως η δημοκρατική, γιατί οι δημοκρατικοί θέλουν και το αντιλαμβάνομαι, το συμμερίζομαι γιατί και εγώ δημοκρατική είμαι. Θέλουν περισσότερες ε, επιβεβαιώσεις για θέματα όπως οι προδιαγραφές για παράδειγμα. Οπότε καλό θα ήταν, ε, αν θέλετε πρόοδο εκεί, να προσετεριστείτε τα μέλη του Κογκρέσου. Για την Κορέα πιστεύω ότι καλό θα ήταν να συνευθεί συμφωνία με τη χώρα αυτή, γιατί αργήσαμε να εξετάσουμε τέτοιες συμφωνίες ε, ελευθέρου εμπορίου με ασιατικές χώρες. Η δική μου έκθεση ψηφίστηκε το 2002. Ήταν σαφές από τότε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπέρ ε, συμφωνιών ελευθέρου εμπορίου με ασιατικές χώρες. Υπήρξαν όμως κάποιες δυσκολίες και ο Ρόμπερτ επισήμανε μία για τους δασμούς. Εγώ έχω μία άλλη που αφορά τους ε, κανόνες προέλευσης τη ρήτρα για την απόσυρση των δεσμών. και το θέμα της προέλευσης είναι πολύ σημαντικό γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση απέρριψε τις συμφωνίες με τις περισσότερες αναπτυσσόμενες χώρες για αυτό το λόγο. Στην περίπτωση της Κορέας τι διαφορές υπάρχουν. Δεν είμαι κατά. Απλώς έχω αμφιβολίες αν είναι καλή συμφωνία, αν είναι επίκαιρη δεδομένου του εργασιακού καθεστώτος εκεί και των προβλημάτων που έχουν οι εταιρείε μα και δεδομένη τη χρηματοπιστωτική κρίση και τη δινή οικονομική κατάσταση, είναι κατάλληλη στιγμή για τη σύναψη μια τέτοια συμφωνία εμπορίου. Αυτή είναι η δική μου προβληματισμή και είμαι ανοιχτή για τη συζήτηση. Πάντως όλα αυτά τα θέματα τα επισημάναμε, αλλά είναι ρητορικά ερωτήματα προς το παρόν δεν έχουν ε, απάντηση. Το θέσαμε και στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την περασμένη φορά. Περιμένουμε τις απαντήσεις ε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το διακανονισμό των διαφορών. Υπήρξε κάποια πρόοδος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη συνάντηση στην Πράγα πριν από δύο εβδομάδες για το Διατλαντικό Κοινοβουλευτικό Διάλογο. Υπήρξε πρόοδος και στο θέμα των ε, των τυχερών παιχνιδιών. Ο Σέλι Μπέκλι που είναι συμπρόεδρος ε, του Διατλαντικού Κοινοβουλευτικού Διαλόγου ε, υποστηρίξαμε και την πρόταση του Γερουσιαστή ΚΟΕΝ. Μάλιστα μας συμπεριέλαβε και στην ιστοσελίδα του. Είπε ότι καταλήξαμε στη συμφωνία για τα θέματα των τυχερών παιχνιδιών του τζόγου και θα δούμε πώς θα δοθεί κάποια συνέχεια. Και χθε έστειλε επιστολή στον κύριο Φερχόγγεν ζητώντα αυτό το θέμα να συμπεριληφθεί στην επόμενη συνάντηση που θα γίνει τον Ιούνιο. Στον επόμενο διακοινοβουλευτικό διατλαντικό διάλογο. Επίσης, ε, σας ευχαριστώ θερμά για την Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης με την ακτή του Ελεφαντοστού. Είμαι ευγνώμων για τις προσπάθειές σας και για την ε, προθυμεί και την ετοιμότητά σας να ασχοληθείτε με τα πιο ακαθόδη ζητήματα. Και αυτό είναι πολύ χρήσιμο και σημαντικό όχι μόνο για μας αλλά και για τις ενδιαφερόμενες χώρες. Συγχαρητήρια. Υποσχέθηκα στους ενδιαφερόμενους ε, στην ακτή του Ελεφαντοστού να κάνω ό,τι μπορώ για να τους βοηθήσω για τα θέματα της τεχνικής αρρωγής και είπα ότι θα κάνω διάβημα και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Απευθύνω έκκληση λοιπόν προς εσάς. Χρειαζόμαστε τη συνδρομή σας. Αν θα μπορούσατε να στείλετε κάποιον εμπειρογνώμονά σας εκεί, θα βοηθήσει πάρα πολύ τους ενδιαφερόμενους στην ακτή του ελεφαντοστού. Το υποσχέθηκα στον κλάδο και γι' αυτό θέλω να τηρήσω την υπόσχεσή μου. Ευχαριστώ πολύ. Στα γερμανικά, Υπάρχει μια ε, παροιμία που λέει ξύπα δεν υπάρχει, όταν δεσμεύεσαι για κάτι το τηρείς». Ε, μας το έχει υποσχεθεί και δεν καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Ε, έχω ακόμα τρεις συναδελφούς που ζήτησαν το λόγο. Θα παρακαλούσα να ακούσουμε ε, και τους υπολείπους και μετά να απαντήσετε. Κύριε Σπορτ, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι τηλεγραφικός. Τι συμβαίνει με την Κολομβία γιατί πριν από λίγο συζητήσαμε το θέμα με έναν γερουσιαστή της Κολομβίας και υπήρξαν βάσιμες αιτιάσεις για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το διαρευνάτε? Μπορεί να μην καταλήξετε σε συμπέρασμα, αλλά ε, θα διερευνηθούν όλες αυτές οι αιτιάσεις και οι καταγγελίες που έγιναν. Γιατί τέτοιες καταγγελίες είχαμε και από το Γενικό Γραμματέα της ε, ETUC. Πιστεύω ότι η διαπραγματεύση αυτή τη στιγμή ε, είναι σε πολύ προχωρημένο στάδιο. Υπάρχουν ορισμένες χώρες που είναι υπέρ των διαπραγματεύσεων, άλλες που είναι υπέρ αλλά δεν είναι ικανές και άλλες που δεν είναι καν πρόθυμες. Εμείς θα είμαστε υπέρ αυτών των διαπραγματεύσεων, αλλά χρειαζόμαστε ένα πλαίσιο για να μπορέσουν και όσοι δεν συμπεριλαμβάνονται ακόμη συμφωνίες να προσχωρήσουν αργότερα. Αποφύγατε έντεχνα να αναφέρετε την Ιαπωνία και την Κίνα, που είναι πραγματικά μεγαθύρια στο παγκόσμιο προσκήνιο, με πολλές διαφορές, αλλά με τεράστια ισχύ. Θα επισκεφτείτε για παράδειγμα την Κίνα. Είναι στο πρόγραμμά σας ε, για τους επόμενους μήνες. Είναι πολύ σημαντικό. Και επανέρχομαι στη Δημοκρατία της Κορέας. Ο Ντέιβιτ Μάρτιν που δυστυχώς απουσιάζει μου ζήτησε να σας το επισημάνω και επισκέφθηκα το Πεκίνο και τη Σεούλ σε πρόσφατη επίσκεψη αντιπροσωπείας ε, της Κορέας και συναντήσαμε τον Υπουργό Εξωτερικών και Εμπορίου στη Σεούλ και είχαμε μια ανταλλαγή απόψεων. Έχω την αίσθηση ότι υπάρχουν κάποιες απόπειρες εκφοβισμού από τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία. Σίγουρα θα υπάρξει κάποιο τίμημα και κάποιο κόστος, γιατί υπάρχουν και ωφέλη. Και μάλιστα τα ωφέλη ε, ξεπερνούν σε μεγάλο βαθμό το τίμημα και τις δαπάνες. Άλλωστε, εξαρτάται από το μέγεθος των αυτοκινήτων ε, που εντάσσεται στη συμφωνία. Αλλά το όφελος θα ξεπεράσει σίγουρα το κόστος. Και το θέμα είναι ότι περιορίζονται στο κόστος και το μεγεθύνουν, ενώ και κάνουν τις προβολές ε, ε, σήμερα για μια κατάσταση που θα λάβει χώρα μετά από πολλά χρόνια. Σε ό,τι αφορά το, το δεσμολογικό καθεστώς, από ό,τι ξέρω είναι ότι οι Κορεάτες είναι υπέρ ε, της ε, πρόοδου, αλλά όχι και υπέρ της κατάργησης. Τι γίνεται όταν αγοράσει κανείς ένα κινητό από την Κίνα και βάζει απλώς μια ετικέτα νοτιοκορεάτικη. Νομίζω ότι εκεί τα πράγματα θα είναι πιο περίπλοκα. Επίση αυτό που με προβληματίζει είναι ότι δεν υπογράψουμε τη συμφωνία με την δημοκρατία της Κορέας. Τι άλλο μας μένει. Δεν υπάρχουν άλλες εναλλακτικέ. Πιστεύω ότι από τη συμφωνία αυτή θα υποφεληθούν και οι δύο πλευρές. Οπότε καλό θα ήταν να δώσουμε έμφαση και να δώσουμε φωνή και σε αυτού που ε, τάσσονται υπέρ των ε, θετικό σημείο και να μην ακούμε μόνο αυτούς που καταδικάζουν αυτή τη συμφωνία. Δεν μπορούμε να ακούμε μόνο αυτούς που προσπαθούν να μας φοβήσουν εξαιτία του κόστους αυτής της συμφωνίας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Καμάλ. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ και την Επίτροπο. Συμφωνώ με πολλά από τα σχόλια που ακούσαμε Μακάρι θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε με τους ε, ε, ε, συμπατριώτες μας, αλλά μια και ανήκουμε σε διαφορετικές πολιτικές οικογένειες, αν εμείς κάνουμε διαβήματα, μάλλον ει βάρο θα είναι. Θα ήθελα να ρωτήσω τις αρχικές σας εντυπώσεις από την ΠΟΕ και μετά τη συνάντηση με την Αμερικανική Αντιπροσωπεία. Εμείς διαπιστώσαμε υπάρχει, ότι υπάρχει μια ένταση μεταξύ των δημοκρατικών στο Κογκρέσο και των δημοκρατικών στην κυβέρνηση. Όταν πήγαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες ε, την εποχή των εκλογών, μίλησα με κάποιους συμβούλους ε, για το εμπόριο και αυτοί που ήταν υπέρ του ελεύθερου εμπορίου από το πλευρό των δημοκρατικών είπαν ότι στο Κογκρέσο υπήρχαν αρκετές εντάσεις. Ποια είναι η δική σας γνώμη. Ακόμη και μετά τις ε, εκλογές στην Ινδία και τη δέσμευσή τους, από τους Αμερικανούς τι δέσμευση έχουμε. Θα μπορέσουμε να ξαναφέρουμε στο σωστό δρόμο της διαπραγματεύσης γιατί έχουν εκτραπεί τον τελευταίο καιρό στην ΠΟΕ. Τι γίνεται με την Ινδία τώρα. Πότε θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις. Βέβαια, ίσως χρειαστεί καιρός για να εξομαλυνθούν τα πράγματα μετά τις εκλογές. από πλευρά μα δεν υπάρχουν αλλαγέ. Και με την Νότιο Κορέα. Συνήθω έχω επιφυλάξει απέναντι σε κλήσει των βιομηχανικών κλάδων. Η αυτοκινητοβιομηχανία στη δεκαετία του 80 και του 90 ήταν κατά των Ιαπώνων λόγω των δεσμολογικών φραγμών. Αλλά τότε δεν ήταν θέμα δοσμολογικών φραγμών, περισσότερο ήταν προδιαγραφών τη Ιαπωνική αγορά. Αυτό που λένε όμω σήμερα οι αυτοκινητοβιομηχανοί είναι ότι θα πρέπει, ε, παρόλο που συμμορφώνονται με τις διεθνείς προδιαγραφές για να ενταχθούν στην, ε, ε, για να προσχωρήσουν στην κορεατική αγορά θα πρέπει να εκπληρώσουν μια νέα σειρά προδιαγραφών. Εγώ δεν θέλω να πηχήσω τις εκκλήσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας, αλλά το θέμα είναι να έχουμε συνθήκες θεμητού ανταγωνισμού και ισοτιμίας. Τώρα για τη συμφωνία με την κοινότητα των Άνδεων. Όταν υπάρχουν πολιτικές διαφορές μεταξύ των διαφορών χωρών και όταν τα κυβερνώντα κόμματα είναι σε διαφορετικά σημεία του πολιτικού φάσματος, υπάρχει μια τάση αυτές οι διαφορές να μεταφέρονται και στις διεθνείς διαπραγματεύσεις. Για παράδειγμα υπάρχουν ισχυρισμοί για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ορισμένες λατινοαμερικανικές χώρες. Η Κολομβία έχει αρκετά προβλήματα Παρ' όλα αυτά, η πρόοδο που έχουν επιτελέσει πολλές χώρες σε σύντομο χρονικό διάστημα είναι αξιοσημείωτη. Μερικοί δεν θέλουν καν βέβαια τέτοια συμφωνία ελευθέρου εμπορίου. Τι θα γίνει όμως η ελήψη μιας τέτοιας συμφωνίας στην Κολομβία και πώς θα αλλάξουν οι σχέσεις της χώρας αυτής με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε περίπτωση μη υπογραφής συμφωνίας. Ευχαριστώ. Ε, κυρία παρακαλώ, το λόγο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να συγχαρώ την αρμόδια επίτροπο για τις άοκνες προσπάθειές της να επιλύσει τα πολυάριθμα προβλήματα του παγκόσμιου εμπορίου και σας εύχομαι καλή επιτυχία και για το δεύτερο μισό της θητείας σας. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε ένα άλλο θέμα. Στα μέτρα κατά του ντάμπινγκ και στην ε, πολιτική αντιντάμπινγκ. Το θέμα αυτό σχετίζεται με την ποιότητα των εισαγόμενων προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρα με το ίδιο το βιωτικό μας επίπεδο και την ποιότητα της ζωής μας. Επίσης είναι ένα θέμα συναφές και με το περιβάλλον. Στην πατρίδα μου τη Βουλγαρία εισάγουμε εδώ και καιρό τοξικό τσιμέντο από γειτονική χώρα, την Τουρκία συγκεκριμένα. Το τσιμέντο αυτό, το σκελοτόμο αυτό, εισάγεται μάλιστα στη Βουλγαρία σε πολύ χαμηλές τιμές, που είναι εμφανώς τιμές dumping. Κάτι τέτοιο οδήγησε στην ε, μείωση της παραγωγής στη Βουλγαρία. Τα μέτρα αντι-dumping θα πρέπει να εξασφαλίζουν προστασία και των παραγωγών αλλά και των καταναλωτών. Ταυτόχρονα θα πρέπει να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ των αντικρώμενων συμφερόντων, ώστε τα μέτρα αντι-dumping να μην ε, γίνουν ένα άλοθη της ε, πολιτικής προστατευτισμού. Κύριε Επίτροπε, ποιο είναι το μακρόπνο όραμά σας για τις πολιτικές αντι-dumping και πιστεύω ότι υπάρχει κίνδυνο στα μέτρα αντι-dumping να μεταμορφωθούν σε μέτρα προστατευτισμού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η Επίτροπος έχει το λόγο, μακρύς ο κατάλογος, Ευρία η παλέτα των ερωτημάτων. Έχετε το λόγο λοιπόν για να απαντήσετε σε όλα αυτά που σας είπα έβαλαν συνάδελφοι. Καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για τα καλά σας λόγια, για μένα και το μέλλον μου. Και ε, όλα αυτά που μου είπατε που θα διαβάσετε στον Πρωθυπουργό μας πραγματικά είναι ευπρόσδεκτα, από όπου και αν προέρχονται. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, εκτιμώ πάρα πολύ αυτά που μου λέτε. Καλωσύνη σας. Λοιπόν, Ρόπερτ, να ξεκινήσω από σένα. Αν επιβεβαιωθεί ο Πασκάλ Λαμή. Ελπίζω ε, να ε, του μιλήσω. Ε, γύρω στις 3 θα το γνωρίζουμε και όλοι παρακολουθούμε τα τηλεγραφήματα και τα νέα. Κατανοώ ότι θα πρέπει να υπάρξει συνέχεια σε αυτή τη δύσκολη χρονική και οικονομική συγκυρία και ο Πασκάλ πραγματικά είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να προωθήσει τη δουλειά στον ΠΟΕ και ιδιαίτερα το γύρο της Ντόχα. Ε, αρχίζω από αυτό που είπατε για την Νότια Κορέα και οι υπόλοιποι και πού βρισκόμαστε με την Νότια Κορέα. Ε, επιτρέψτε μου να βάλω λίγο ένα ιστορικό πλαίσιο εδώ και υπόβαθρο. Πρώτον, εγώ δεν ενδιαφέρομαι να κάνουμε μια συμφωνία που να μην είναι υπέρ ε, της Ένωσης και σε πολύ μεγάλο βαθμό των, επι, των επιχειρήσεων. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα κοιτάμε τι προσθέτει μια συμφωνία και τι προσφέρει ε, στη βιομηχανία μας. Επιπλέον η αυτοκινητοβιομηχανία ε, θέλει οπωσδήποτε να φροντίσουμε ε, ό,τι κάνουμε να είναι προς όφελός του στο μέλλον και ό,τι κάνω εγώ προσωπικά. Εγώ δεν πιστεύω ότι η συμφωνία αυτή θα σημάνει το τέλος της αυτοκινητοβιομηχανίας ούτε ότι αυτή καθ' αυτή η αυτοκινητοβιομηχανία θα πάρει την κατιούσα τώρα οικονομικά. Είναι καλή συμφωνία. Αυτό είναι δικό μου μέλημα και για την οικονομία και για τα αυτοκίνητα. Πριν από δύο χρόνια που ξεκινήσαμε, ε, πολλοί συνάδελφοι άρχισαν να συνεργάζονται ακριβώ με τον κλάδο. Ο, ο, ο κύριος Καμάλ ε, μίλησε κυρίω για εμπόδια μη, μη ε, δασμολογικά, προδιαγραφές και πρότυπα κτλ. Ασχοληθήκαμε με το καθένα ξεχωριστά. Και τώρα μέσα στη συμφωνία καταφέραμε να πετύχουμε να συνεχιστούν οι εξαγωγέ μας. Είναι 3% βέβαια η συμμετοχή μα ε, στην Νότια Κορέα. Το μερίδιο του είναι μεγαλύτερο. Και θέλουμε να διευρεθεί το δικό μα. Ορισμένοι κατασκευαστέ έλεγαν, α πούμε, «Ε, οι Κορεάτε έχουν στάνταρ Καλιφόρνια. Εμεί που στέλνουμε αυτοκίνητα στην Καλιφόρνια με τι ίδιε προδιαγραφέ μπορούμε να στείλουμε και στην Νότια Κορέα. Είναι μεγάλο το κόστος, αλλά δεν είναι ανυπέρβλητο. Έτσι, όλα αυτά χρειάστηκε να τα λύσουμε. Θα είναι ανοιχτή αγορά λοιπόν για τους κατασκευαστές μας. Και υπάρχει αγορά. Για μικρά αυτοκίνητα ε, premium πήγα στην Κορέα και επισκέφθηκα το εργοστάσιο της Ρενό που έχει εργοστάσιο στην Κορέα Ρενό για να δω τι κάνει. Ε, είμαι λοιπόν αρκετά πεπισμένη ότι το αναγνωρίζει αυτό βιομηχανία αυτό προσπάθεια και το, και το πράττει. Υπάρχει επίση μια γνήσια ανησυχία από πλευρά τη αυτοκινητοβιομηχανία για τον τρόπο με τον οποίο θα του επηρεάσει η συμφωνία αυτή ε, ω προ την ικανότητά του να διατηρήσουν το μερίδιο αγορά. Να σα δώσω μερικά στοιχεία και πάλι να αναφεσπίτητε. έτσι. Ε, υπάρχει μια δυνατότητα, πιστεύουμε, 650 κορεατικά αυτοκίνητα να απορροφηθούν στην Ευρώπη πριν την ύφεση. 600.000 αυτοκίνητα φέτος κορεατικά ε, θα κατασκευαστούν στην Ευρώπη και δημιουργούνται εκεί θέσει απασχόληση. Θαυμάσια, καταπληκτικά. Λοιπόν, είναι περιθωριακό ο αντίκτυπο, 50.000 περίπου δηλαδή. Και σύμφωνα με πληροφορίε που έχουμε, οι καταναλωτέ επιλέγουν μεταξύ κορεατικών και ιαπωνικών. Δηλαδή, ε, δεν είναι ανταγωνιστικά τα κορεατικά αυτοκίνητα προς τα ευρωπαϊκά, προς τα ιαπωνικά είναι. Ακόμα και συνέβαινε αυτό το θεωρητικό, ας το δεχτώ ενδεχόμενο, μιλάμε για μια κατάσταση όπου η Κορέα ήδη κατασκευάζει εδώ αυτοκίνητα. Δηλαδή, είναι εδώ τα αυτοκίνητα, δεν θα έρθουμε τη συμφωνία. Δεν βάζουμε κάποιους φραγμούς για να μην μπουν. Κατασκευάζονται εδώ. Το θέμα είναι τώρα πώς υποστηρίζει κανείς μια οικονομική συμφωνία που από τη μια θα αλλάξει το μέλλον της αυτοκινητοβιομηχανίας, δηλαδή ε, θα βάλουμε καλύτερο πλαίσιο και οικονομικές συνθήκες ε, για την εγχώρια αγορά. Είναι εγχώρια αγορά αυτοκινήτων. Έτσι θα βοηθήσουμε τον κλάδο να ορθοποδήσει. Γιατί όλοι εμείς αγοράζουμε για νεωρία αυτοκίνητα. Καλά, εξάγουμε κιόλα, αλλά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τις εξαγωγές. Λοιπόν, θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι θα έχουμε πραγματικές ευκαιρίες όσο γίνεται για περισσότερους κλάδους της οικονομίας. Ε, και επίσης έμεσα υποστηρίζουμε και άλλους κλάδους της ε, βιομηχανίας αλλά και τα αυτοκίνητα. Λοιπόν, θα σας έλεγα ότι αυτό που έχουμε τώρα θα έρθω σε λίγο στο ιδιαίτερο που ρωτήσατε. Ε, το έχουμε διαπραγματευτεί πάρα πολύ προσεκτικά. Βέβαια, οι εκτιμήσεις ποικίλουν, αλλά μιλάμε για 20 δισεκατομμύρια οικονομική ανάπτυξη. Ορισμένες χώρες έχουν κάνει υψηλότερε εκτιμήσει, η Γερμανία, δεν θα το πω εγώ αυτό, αλλά η γερμανική κυβέρνηση. Πάντως μιλάμε για δισεκατομμύρια ευρώ. Χημική βιομηχανία, υπηρεσίε, ε, ε, μηχανική, ε, φαρμακευτικά προϊόντα. Μεγάλο κέρδος λοιπόν θα είναι για τις οικονομίε Ευρώπης και μεταξύ αυτών και την αυτοκινητοβιομηχανία. Το ειδικό πρόβλημα που αφορά τα αυτοκίνητα είναι ε, η παναχώρηση, η drawback. Ε, πρόσφατα στο Λονδίνο μου είπαν οι κοράτες ότι είναι εγώ έγινε γραμμή για εκείνους. Όχι για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά ξεκαθάρισαν ότι και αυτό είναι πάντα επιχείρημα για καλύτερη συμφωνία, ότι υπάρχει πρόβλημα. Δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα οι διαπραγματεύσεις, ούτε πρόκειται να σας αποκαλύψω πάρα πολύ τα χαρτιά μου, αλλά συμφωνώ με αυτό που λέει και ο Γκλίν Φόρτ, ότι επιθυμεί η κορεατική κυβέρνηση να συναυθεί αυτή η συμφωνία και ο Υπουργός Κιμ, Κιμ ε, όντως ενδιαφέρεται πάρα πολύ. 150 εκατομμύρια ευρώ δεχομένω. Ε, αλλά μιλάμε για τις εκατομμύρια που θα εισρέψουν. Δηλαδή είναι τα ανταλλάγματα προφανώς που δίνει κανείς σε τέτοιες περιπτώσεις. Τα αντισταθμιστικά. Το βασικό τώρα ερώτημα είναι πώς θα βεβαιωθούμε ότι δεν θα υπάρξει αυτό το τριγωνικό εμπόριο, να εισάγουν κάτι από την Κίνα, να βάλουν κορεατική ετικέτα και να το εξάγουν. Μα υπάρχουν οι κανόνες για την προέλευση, είναι σημαντικά αυτά τα θέματα και διέπουν τις συμφωνίες για να βεβαιωθούμε ακριβώς ότι δεν θα έχουμε κορεατικοποίηση κινέζικων προϊόντων. Υπάρχουν όμως και Ευρωπαίοι κατασκευαστές που παράγουν στην Κορέα και εισάγουν εξαρτήματα και ανταλλακτικά από τρίτες χώρες. Προσοχή να μην σκοτώσουμε και την ευρωπαϊκή βιομηχανία εκεί. Γιατί πολλέ πρώτε ύλε δεν τι βρίσκουν επί τόπου, αλλά τι εισάγουν από αλλού. Ευρωπαϊκέ εταιρείε, επαναλαμβάνω, στην Κορέα. Και αυτό θα πρέπει να το σκεφτούμε. Πάντως έχουμε το συνδυασμό των κανόνων προέλευση και το γεγονό ότι το προϊόν θα πρέπει εν μέρη να κατασκευάσετε στη Γορέα. Ποιο μέρο τώρα θα κατασκευαστεί και αυτό είναι αντικείμενο ακόμα διαπραγμάτευση. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά. Λοιπόν, σα στέλνω το εξή μήνυμα. Έχω υπόψη μου πάρα πολύ καλά τα μελήματα της αυτοκινητοβιομηχανία. του έχω συναντήσει, γνωρίζουν ότι η πόρτα μου είναι ανοιχτή. Θα χρειαστούν 5-6 χρόνια ακόμα με την καλύτερη βούληση όλων για να εφαρμοστεί η ε, συμφωνία και μέχρι τότε ελπίζουμε να έχουμε ξεπεράσει την ύφεση και να επανέλθει η οικονομική μεγέθυνση. Αλλά πολλά πράγματα είναι επωφελή για μας και ευεργετικά. Είναι μεγάλη αγορά. Και από την αρχή θα ανοίξει για μας. Αυτό είναι πάρα πολύ καλή συμφωνία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έρχεται σε περιόδους πραγματικά πολύ δύσκολες για την οικονομία μας, με μεγάλο άγχος και πίεση και έτσι θα αποφεληθούν οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες, αλλά να δούμε με ποιο τρόπο θα ληφθεί υπόψη ακριβώς αυτός ο ευάλωτος χαρακτήρας της αυτοκινητοβιομηχανίας. Δεν θέλουμε να τους υπονομεύσουμε. Τις ευκαιρίες τους θέλουμε να αυξήσουμε. Και σας λέω, τα καωριατικά αυτοκίνητα ήδη κατασκευάζονται στην Ευρώπη. Εμεί δεν έχουμε κανένα μοχλό ούτε κανένα όφελος εμπορικό. Η ευκαιρία λοιπόν είναι να χρησιμοποιήσουμε το εμπορικό αυτό μέσο πίεση και να μην το απεμπολίσουμε. Δεύτερον, Πολλοί συνάδελφοι το έθεσαν αυτό και είναι η Αμερική και ο γέρος της Δόχα. Πήγα στο Κογκρέσο όπως και η Έρικα Μάν και άλλοι. Μίλησα με τους κατασκευαστές, μίλησα με τους αγρότες, με τα συνδικάτα. Το ε, προέδρους διαφόρων επιτροπών, Ways and Means ε, του Κογκρέσου και άλλων που ασχολούνται με θέματα εμπορίου, με ερωτήσεις, απαντήσεις και επαφές διάφορες. Έχεις απόλυτο δίκιο, Έρικα. Είναι τεράστιο αυτό το θέμα. Το Κογκρέσο θεωρεί αυτό το θέμα θετικό για τις Ηνωμένε Πολιτείε. Αν αρχίσουμε τώρα να ξυλώνουμε όλα τα θέματα που είναι επιτάπητος, δεν πρόκειται να προχωρήσει εκπρόσωπος τον είπα ε, στο εμπόριο θέλει λέει να αξιολογήσει το, το καθεστώς που ισχύει, τι σημαίνει αυτό για την Αμερική, τι ε, ευεργετήματα έχουν και πώς μπορούν να προχωρήσουν. Τώρα για τους Αμερικανούς, αυτό που έχει σημασία είναι να περιορίσουν λίγο ε, τις ε, προσδοκίες που έχουν από τις αναπτυσσόμενες και αναδυόμενες χώρες. γιατί θεωρούν ότι οι χώρε αυτές αμασάνε λίγο τα λόγια τους. Ε, υπάρχει ο στόχο 30%, ζήτησαν 6 μήνε να το σκεφτούν. Εγώ έχω την εντύπωση ότι κινούνται γρηγορότερα. Πάντως στο τέλος ο Λευκός Οίκο παίρνει την πολιτική απόφαση και το Κογκρέσο ακολουθεί είναι σημαντικό να αποφασίσουν να επιστρέψουν στο γύρο της Δόχας. Θα δούμε τι θα γίνει και με τις διμερείς συμφωνίες που συζητούν. Πάντως είναι δύσκολη η κατάσταση γιατί πολλές κατασκευαστικές, μάλλον εργοστάσια, ε, γεωργοί ανησυχούν, ανησυχούν από ότι στο παρελθόν περισσότερο Υπάρχουν δυσκολίες. Συνεχίζω σύντομα. σε άλλα θέματα που έθεσε η Έρεκα. Α, για τα τυχερά παιχνίδια. Ξέρετε ότι έχω κάνει μια έκθεση, να δούμε τι θα βγει. Ε, σας ευχαριστώ πολύ. Ναι. Για την ακτή ελεφαντοστού βεβαίως θα σας υποστηρίξουμε σε ό,τι χρειάζεστε και θα είναι στη διάθεσή σας οι συνάδελφοι από τις υπηρεσίες μας. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι η υπογραφή συμφωνίας σηματοδοτεί την αφετηρία και όχι το τέρμα μιας προσπάθειας ε, σε οικονομικούς και εμπορικούς όρους. Γκλίν Φόρτ ε, μου έθεσε διάφορα ζητήματα. Θα προσπαθήσω να απαντήσω. Και για την Κολομβία που είπε σε παρόδο. Με μεγάλη προσοχή κοιτάμε τι λένε τα Ηνωμένα Έθνη και ο Διεθνή Οργανισμό Απασχόληση, το Διεθνέ Γραφείο Απασχόληση. Βεβαίω ανησυχούμε, το είπε και εσύ. Υπάρχουν στοιχεία γι' αυτό. Στο μεταξύ όμω προ το παρόν Μπορεί να ανησυχούμε, αλλά δεν είμαστε στο στάδιο να ζητήσουμε έρευνες επίσημες και ε, ανακρίσεις, ας πούμε, για να δούμε τι γίνεται. Μπορεί να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Εγώ τι θέλω με κάποια άλλα κράτη. Να θεωρήσουμε, νομίζω το έχω ξαναπεί στην Επιτροπή σας, ότι το εμπόριο είναι ε, μία ψηφίδα σε ένα ολόκληρο ψηφιδωτό. Δεν διέπεται το σύνορο των σχέσεων με της Ευρωπαϊκής με άλλα κράτη από το εμπόριο. Και δεν μπορεί παρά να είναι ένα κομματάκι του πάζελ το εμπόριο. Δεν στέκει από μόνο του. Υπάρχει ένα σύνολο σχέσεων. Θα πρέπει λοιπόν να ξέρουμε ότι στις γενικές σχέσεις που έχουμε ε, αντιμετωπίζουμε και το εμπόριο. Το γνωρίζει ο Υπουργός της ε, Κολομβίας. Πέρσι συναντήθηκα με τον Πρόεδρο πριν γίνω Επίτροπος. Είναι πραγματικά συναρπαστικό να δει κανεί τι αλλαγές έχουν γίνει στην Κολομβία είναι προ όφελο τη Κολομβία και εναπόκειται σε εσά να το αποδείξετε αυτό. Θα πρέπει να συνεχίσουμε προ την κατάσταση αυτή, να σταματήσουν να τερματιστούν τελείω οι παραβιάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μετά να συνεχίσουμε. Βεβαίω θα έχω υπόψη μου όλα αυτά και τα γνωρίζω. Τώρα, για τι χώρε ΑΣΕΑΝ, Νοτιοανατολική Ασία. Συμφωνώ. Βιετνάμ, Σιγκαπούρη, ενδεχομένω η Ταϊλάνδη είναι τρει χώρε που μάλλον θα προχωρήσουν περισσότερο και εύχομαι και ελπίζω να γίνει αυτό για την Κίνα. Έρχεται την άλλη εβδομάδα ο αντιπρόεδρος κινέζικης κυβέρνησης για να ε, προεδρεύσει μαζί μου ε, σε ένα διάλογο υψηλού επίπεδου και θα έρθουν καμιά ε, 10 με 12 υπουργοί μαζί του και με την Επιτροπή θα συζητήσουμε διάφορα θέματα, εμπόριο, επενδύσεις και άλλα, επιχειρήσεις κτλ από διάφορες ε, σκοπιές, από διάφορα χαρτοφυλάκια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα έχουμε και ένα γεύμα με μεγάλους διευθυντές επιχειρήσεων, ε, εκτελεστικούς διευθυντές ευρωπαϊκών επιχειρήσεων για να δούμε πώς θα επανέλθουμε το Σεπτέμβριο. Και θα ανταποδώσω εγώ αυτή την επίσημη επίσκεψη. Για την Ιαπωνία. Γνωρίζετε ότι προσεχώς θα έχουμε στην Πράγα τη Σύνοδο Κορυφής Ιαπωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θα ήθελα να μπω αυτή τη στιγμή σε αυτό το θέμα. Αργότερα θα τα ξαναπούμε. Με τα θέματα πολέμηση του ντάμπινγκ, έτσι, νομίζω είναι το μόνο που εκκρεμεί ακόμα σε απάντηση. Προς την κυρία Λούπτσεβά, από τη Βουλγαρία, σωστά το λέω, ναι. Το αντι είναι πραγματικά ένα θέμα αποκαλύπτει ένα φάσμα απόψεων. Ε, η δική μου άποψη λέει ότι υπάρχουν κάποιοι κανόνες και θα πρέπει να τους εφαρμόσουμε. Και στην παρούσα οικονομική συγκυρία θα πρέπει να εφαρμόζονται ε, νομότυπα, ε, σχολαστικά και με ειλικρίνεια. Καταλαβαίνω ότι αυτό τον καιρό η βιομηχανία μας είναι πιο ευάλωτη στο ντάμπινγκ και χρειάζεται να δράσουμε. Πέφτουν και οι τιμές όμως γενικά. Αυτό θα πρέπει να δούμε τι είναι dumping και τι δεν είναι. Έτσι. Εξαρτάται από το πώς τη θεώρηση έχουμε. Μάκρο πρόθεσμα τώρα. Πρέπει να γίνει μια συζήτηση πιστεύω. Γιατί εδώ και καιρό εκρεμεί. Ε, η γενική ιδέα είναι πώς θα βεβαιωθούμε ότι αυτά που κάνουμε αποσκοπούν γνήσια στο να τερματιστούν οι κακές πρακτικές για να υποστηρίξουμε στο μέλλον τις επιχειρήσεις μας να έχουν το μερίδιο αγοράς τους και δεν θέλουμε να είμαστε προστατευτιστές. Είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να προστατεύουμε την οικονομία μας από τον ντάμπινγκ και η πρώτη δική μου δουλειά είναι να υποστηρίζω την ευρωπαϊκή οικονομία. Νομίζω ότι τα κάλυψα όλα. Ζητώ συγγνώμη αν ξέχασα κάτι. Ελπίζω να σας καλύψουν αυτά, να είπα αρκετά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Απαντήθηκαν οι ερωτήσεις. Έβλεπα τους συναδέλφους να ανέβουν καταφατικά από πάνω προς τα κάτω. Και η κυρία Λούπτσεβα είναι δεξιά, από δεξιά προς τα αριστερά όταν ε, θέλει να πει ναι στη Βουλγαρία. Ελοκληρώνονται εδώ οι εργασίες της Επιτροπής μας. Έχουμε μια μικρή δεξίωση από χαιρετιστήρια ετοιμάσει. Παρακαλώ να βγούμε έξω για λίγο να παραμείνουν λίγο οι συντονιστέ. Ένα λεπτάκι, πολύ σύντομα θα κάνουμε μια επίσημη συνεδρίαση των συντονιστών. Όλοι οι υπόλοιποι είστε ελεύθεροι. Παρακαλώ. Ερχόμαστε αμέσω. Αφήστε την πόρτα για μα. Ευχαριστώ. Κανονικά οι συντονιστέ συνεδριάζουν και κλεισμένο των θυρών. Αλλά για να μην αργήσουμε, σα κάνω την εξή πρόταση. Έχετε λάβει τα σημειώματα που σας έχουν αποσταλεί και ρωτώ τώρα γενικά. Ε, συνολικά οι παρόντες συντονιστές συμφωνούν με όλες τις προτάσεις που έχουν λάβει. Also, Sie Συμφωνείτε με όλες τις προτάσεις. Ωραία. Μπορούν έτσι να γραφτούν αυτά στα πρακτικά Ολοκληρώνω τη συνεδρίαση των συντονιστών. Ευχαριστώ για τις διερμηνεί. Είστε όλοι προσκεκλημένοι στη δεξίωση. Μη μα φύγετε οι διερμηνεί. Βγείτε και πάρτε κάτι να φάτε στο βαθμό που θα σα αφήσουν κάτι. Και επειδή προσωπικά δεν θα ξανάρθω, θέλω να σα ευχαριστήσω όλους. Κάνατε καταπληκτική δουλειά. Η Έρικα. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας ευχαριστήσω εγώ εξ ονόμα της πολιτικής μου ομάδας προσωπικά. Στην αρχή είχαμε κάποιες επιφυλάξεις, δεν είναι πάντα τόσο εύκολα τα πράγματα ε, να έχεις πρόεδρο και να δεχτεί κανείς ένα πρόεδρο από τη δική σας πολιτική παράταξη. Πάντως ήταν όλα πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ ευχάριστα και ελπίζω να μην χαθούμε.